Uh, morning, uh, ladies and gentlemen, uh, welcome Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην πρώτη συνεδρίαση της νέας χρονιάς της Επιτροπής ε, Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Ο Σεφ λοιπόν, καλωσορίζω ιδιαίτερα και τους βοηθούς, τη γραμματεία και τους εισηγητές μας για τα βασικά θέματα που είχαν πολλή δουλειά στις διακοπές γιατί χρειάστηκε να επεξεργαστούν πολλοί άριθμες τροπολογίες. Θα ακούσουμε αργότερα την κυρία Βερνιό και τον κύριο Ζουβά. Καλή χρονιά σας εύχομαι. Ελπίζω να επιστρέψετε ακμαίοι και ανανεωμένοι από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές γιατί μας περιμένει πολύ φόρτος αυτή τη χρονιά. Και άλλωστε είναι και η τελευταία χρονιά πριν το 2014 που θα είναι έτος ευρωεκλογών. Βλέπετε πόσο ραγδαία κυλάει ο χρόνος στην πολιτική. Θα ήθελα να καλωσορίσω και όλους όσους μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο. Ετοιμάζουμε και τον νέο μας έντυπο, το IMCO News, τη νέα έκδοση, αλλά λίγη υπομονή γιατί δεν είναι έτοιμο ακόμα. Σας έχουμε μοιράσει την ημερήσια διάταξη. Να, θεωρώ ότι, ε, μπορούμε να, την, ε, να θεωρήσω ότι μπορούμε να την εγκρίνουμε. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Εγκρίνεται. Ε, υπάρχει ένα ε, θέμα με το διορθωτικό. Μία τεχνική αλλαγή δηλαδή, ένα κορυγκέντουμ στον πρόσφατο κανονισμό για την έγκριση αγροτικών και δασικών οχημάτων. Εκεί αναφέρονται ανακριβώς κάποιες ημερομηνίες το διορθώσαμε με τον εισηγητή κύριο Παντζέρη, το ενέκριναν και οι συντονιστέ. Θα πρέπει όμω να το εγκρίνουμε επίσημα και στην Επιτροπή. Το έχετε λάβει στα δοσιέ σα και αν δεν, υπάρξουν αντιρρήσεις, αν δεν υποβληθούν αντιρρήσει μέχρι το τέλο τη συνεδρίασής μα σήμερα, θα θεωρήσω ότι έχουμε επίσημα εγκρίνει και το διορθωτικό. Περνάμε τώρα σε ένα από τα θέματα που μας απασχολούν κατά προτεραιότητα εδώ και πολλά χρόνια υπό την ηγίδα της κυρίας Βερνιό που είναι η συγγήτρια για την οδηγία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Θα της δώσω το λόγο για να μας σχολιάσει τις συμβαστικές τροπολογίες. Χαίρομαι γιατί είναι παρόντες και οδησηγητές, η κυρία Λαγκρίπ από το ΕΛΚ, η κυρία Παρβάνοβα θα αναπληρώσει τον κύριο Μπουσόη, Τούρινεν από το από τους συντηρητικούς. Κάποιος που απουσιάζει δικαιολογείται. Είναι λοιπόν, έχουμε απαρτία σε ό,τι αφορά το επιτελείο που ασχολείται με το θέμα αυτό και καλωσορίζω και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα μας ενημερώσουν για τις εξελίξεις. Χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν, να δώσω το λόγο στην Περναντέτ Βερνιό, την εισηγητριά μας, για να μας παρουσιάσει τις συμβαστικές τροπολογίες. Έχεις το λόγο, Περναντέτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και πριν να αρχίσουμε με τη συζήτηση θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία, επικοδομητική εργασία και είμαστε από τις σπάνιες ε, επιτροπές κύριε Πρόεδρε που έχουμε τόσο αγαστή συνεργασία μεταξύ των πολιτικών ομάδων και έτσι πραγματικά φαίνεται η κοινοτική υπεραξία και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό και να το τονίζουμε γιατί εργαζόμαστε με βάση κυρίως το κοινοτικό συμφέρον και το γενικό συμφέρον και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί και αυτή συνέβαλε στην αγαστή συνεργασία και ας μην ξεχνούμε και τους διερμηνείς για την δική τους συμβόλη. Καλή χρονιά σας έχουμε λοιπόν και πάλι. Περνάμε τώρα στο θέμα της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Εδώ και μήνες συναντιέμαι τακτικά με τους σκιώδεις ηγητές, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για το έργο τους, προκειμένου να καταλήξουμε στις συμβαστικές τροπολογίες για τα πιο θεμελιώδη ζητήματα αυτής της οδηγίας, Έχοντα υπόψη φυσικά την ανάγκη συμφιλίωση και των διστάμενων απόψεων όπω παρουσιάζονται στι πολυάριθμε τροπολογίε, πάνω από 700, αλλά και συνεχίζοντα το διάλογο με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συμβαστικέ τροπολογίε που θα εξετάσουμε σήμερα και που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, γιατί έχει προγραμματιστεί και μια τελευταία συνεδρίαση με του κοιόδη ηγητέ την επόμενη Τετάρτη, αντικατοπτρίζουν τις βασικές αρχές ε, όλων των πολιτικών ομάδων. Απαναλαμβάνω, τα κείμενα δεν έχουν οριστικοποιηθεί, γιατί την Τετάρτη θα τα ε, συζητήσουμε και θα διευθετήσουμε και τα εκκρεμή ζητήματα πριν ε, αποκρισταλωθεί η τελική του μορφή. Θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε γενική επισκόπηση στα 12 θεμάτων. Σε ό,τι αφορά τη μερική πρόσβαση. Η μερική πρόσβαση θα πρέπει να γίνεται περιπτωσιολογικά, να αποφασίζεται περιπτωσιολογικά και να μπορεί η αρμόδια αρχή να απορρίπτει την μερική πρόσβαση για λόγους ε, δημόσιου συμφέροντος. Θα πρέπει βέβαια ε, τους επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος να τους ορίσουμε στο κείμενο. Κάτι που έγινε με βάση την, τον ορισμό της οδηγίας για τις υπηρεσίες και με παραπομπή στην ομολογία του ΔΕΚ. Επιπλέον προσθέσαμε τρεις όρους για την ε, έγκριση της μερικής πρόσβασης. Μία πλήρη ε, κανονική ε, πρόσβαση έχει απορριφθεί. Δεύτερον, έχουν αναγνωριστεί οι επαγγελματίες στη χώρα προέλευσης και τρίτον, να μην πρόκειται για το μεακό επάγγελμα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ασκήσεις μαθητείας, τα στάζ, σε ό,τι αφορά την αμοιβή αυτών των ε, περίοδων μαθητείας. Έχει καταργηθεί το θέμα της ε, αμοιβή, αλλά διευκρινίζεται ότι η οδηγία εφαρμόζεται μόνο στις μαθητείες που εντάσσονται στη κατάρτιση για ένα κατοχυρωμένο ρυθμισμένο επάγγελμα. Επιπλέον, ε, προβλέψαμε κάποια χέγγια για, τις, για το σεβασμό των εργασιακών συνθηκών στα πλαίσια αυτών των μαθητιών. Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική ταυτότητα. Για την επαγγελματική ταυτότητα επιλέξαμε την εξή λύση. Πίστευα ανέκαθεν ναι, ότι είναι αναγκαίο να διαφυλάξουμε την αρχή της σιωπηρής αναγνώρισης, που είναι το μόνο, ο μόνος τρόπος ε, για να αντιμετωπίσουμε τη δυσφορία και τα παράπονα των επαγγελματιών. Βέβαια θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η σιωπηρή αναγνώριση δεν ισοδυναμεί με δικαίωμα άσκησης θα πρέπει να συνοδευτεί από μια χαλάρωση των προθεσμιών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα μιας περίοδου αναστολής σε περίπτωση αίτησης για συμπληρωματικές πληροφορίες. Η υποχρέωση ενημέρωσης των επαγγελματιών έχουν ε, διευρυνθεί με λογικό τρόπο. Σε ό,τι αφορά το μηχανισμό προειδοποίησης. Όλοι χαιρετίζουμε τον νέο μηχανισμό, αλλά οι τρόποι εφαρμογή του δημιουργούν ακόμη κάποια προβλήματα εξαιτίας κυρίως του γεγονότος της ε, ποικιλομορφίας ε, των αθηνικών νομοθεσιών και του εθνικού δικαίου. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν ε, τις ιδιαιτερότητες αυτές προβλέποντας θέμα παρά του μηχανισμού σε περίπτωση παραποίηση των εγγράφων. Σε ό,τι αφορά τα γλωσσικά θέματα. Υπάρχουν πρακτικά ζητήματα. Θα πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση του επιμερισμού των ευθυνών <clears throat> και ε, για τον έλεγχο είναι μόνο οι αρμόδιες αρχές, η λήψη αυτών, ε, ένας οργανισμός που καθορίζεται από τα κράτη-μέλη. Επιπλέον είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα τεκμήρια αποδείξεις που προσκομίζει ο επαγγελματίας ότι αφορά τη γνώση της γλώσσας και καλό θα να θεσπιστούν κάποια στερεότυπα τεστ με πρότυπο αυτά που υπάρχουν για τις σπουδές στο εξωτερικό. Ένα θέμα που έχει παραμείνει εκρεμές είναι το θέμα των χωρών που έχουν περισσότερες από μία επίσημες γλώσσες. Δεν θέλουμε να υποχρεώσουμε τους επαγγελματίες να μάθουν μια επιπλέον γλώσσα, αν κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο για την ε, άσκηση του επαγγελματός τους. Και εδώ πέρα έχω κατά νου κυρίως στο Βέλγιο. υπάρχει και το θέμα της Ισπανίας και εκεί έχουμε αυτόνομες περιφέρειες όπως η Καταλωνία με δική τους γλώσσα. Το θέμα θα διαθετηθεί την επόμενη Τετάρτη, γιατί επαναλαμβάνω έχει μείνει ανεπίλητο προς το παρόν. Δεν πιστεύω ότι είναι σκόπιμο αυτή τη στιγμή να θεσπίσουμε υποχρέωση ε, για την εκμάθηση μιας περιφερειακής γλώσσας ε, ε, σε χώρες μάλιστα που αντιμετωπίζουν σχετικές πολιτικές δυσκολίε. Τώρα, για την συνεχή ε, κατάρτιση προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ε, ψηλή ποιότητα της περίθαλψης και την υγεία των ασθενών, καθώς και τη διαβίου κατάρτιση, είναι σημαντικό να προβλέψουμε και απαραίτητο να προβλέψουμε μια συνεχή εκπαίδευση για τα ιατρικά επαγγέλματα, τα επαγγέλματα υγείας, υπό την ευθύνη των κρατών μελών που θα πρέπει να μπορούν να ελέγχουν το επίπεδο της ε, επιμόρφωσης αυτής σε ό,τι αφορά το κοινό πεδίο κατάρτισης. Το κοινό αυτό πεδίο είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της πρότασης και συνάδει με το κοινοτικό σχέδιο, γιατί έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε μια μετάβαση προς το ε, μηχανισμό της αυτόματης αναγνώρισης. Θέλουμε να γίνει μια επέκταση στα επαγγέλματα αυτόματης αναγνώρισης ε, φυσικά φροντίζοντας, ε, τις, ε, φροντίζοντας για τη συμμετοχή και των επαγγελματικών οργανώσεων στην κατάρτιση αυτών των μηχανισμών. Σε ό,τι αφορά τα κατοχυρωμένα επαγγέλματα, προτείναμε μία ενημέρωση των απαιτήσεων εκπαίδευσης, αλλά προσπαθήσαμε να διασκεδάσουμε και κάποιες ανησυχίες που εκφράστηκαν. Σε ό,τι αφορά τις βασικές ιατρικές, την βασική ιατρική εκπαίδευση, προτείναμε εξαετή εκπαίδευση με δυνατότητα αναγνώριση εναλλακτική εκπαίδευση πέντε ετού διάρκεια, όπως ισχύει σε ορισμένα κράτη-μέλη. Υπό τον όρο όμως ότι θα τηρούνται οι 5.500 ώρες και λαμβάνονται υπόψη διατάξει του νέου άρθρου 21α. Σε ό,τι αφορά τους οδοντιάτρους, χρήσιμο είναι και υπευλήθησαν πολλές ε, ερωτήσεις σχετικά να γίνει μια ενημέρωση των προσόντων και των δεξιοτήτων ε, των εδοντιάτρων, 5.000 ώρες τουλάχιστον, και μια εναρμόνιση του πεδίου αρμοδιοτήτων τους. Και επίσης θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη τις ιδιαίτερες παθολογίες ε, για τους στοματολόγους και τις ειδικότητες άλλες των οδοντιάτρων. Τώρα, για τις ΜΕΣ Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αυτά τα 12 χρόνια που είναι απαραίτητα ε, και επίσης να διευκρινιστεί ποιο είναι το απαραίτητο πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. Και εκεί ε, φαίνεται ότι καταλήξαμε συμφωνία με το Συμβούλιο για τις ΜΕΣ, κάτι που δεν ήταν προφανές από την αρχή. Για τους φαρμακοποιούς. Και εδώ υπήρχαν εξέλιξεις στο επάγγελμα και το άρθρο 45.2 θα πρέπει να επικαιροποιηθεί, όπως πρότεινε και η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Για τους αρχιτέκτονες υπάρχει γενική υποστήριξη ε, για τη μετάβαση σε μια εξαιτή εκπαίδευση. Βέβαια, για να ληφθούν υπόψη οι διάφορες οργανώσεις ε, των εκπαιδεύσεων, προτάθηκε και τρίτη λύση, προβλέποντας τη δυνατότητα να έχει κανεί ισοδύναμο μια χρονιά πρακτική εκπαίδευση στη διάρκεια των σπουδών, ακόμη και μέσα των σπουδών και όχι μόνο μετά το πέρα του, ώστε να διορθωθούν κάποιε δυσκολίε που αντιμετωπίζουν χώρε όπω η Ισπανία. Γιατί εκεί οι φοιτητέ αρχιτεκτονική ε, δεν μπορούν εύκολα να βρουν στάζ ε, κατά το τέλο των σπουδών του. Ό,τι αφορά του συμβολογράφου και τι ε, νοσηλεύτριε νοσηλευτέ, τα δύο πιο επίμαχα σημεία, για τα δύο επαγγέλματα λοιπόν, οι συζητήσεις είναι περίπλοκες στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά εμείς καταφέρουμε τουλάχιστον να έχουμε οικοδομητικές συζητήσεις, αλλά έχουμε τεράστιες δυσκολίες με το Συμβούλιο για τα δύο αυτά επαγγέλματα. Δεν έχει υποβληθεί ακόμη συμβαστικό κείμενο. Θα το εξετάσουμε Τετάρτη. Αναζητούμε λοιπόν μια λύση για τα δύο αυτά επαγγέλματα, κάτι που θα είναι και η προτεραιότητά μα η και για την επόμενη Τετάρτη, αλλά και για την ψηφοφορία στις 23 Ιανουαρίου. Για τους συμβολογράφους πιστεύω ότι θα καταλήξουμε στη συμφωνία. Για τις νοσηλεύτριες, νοσοκόμους, επαναλαμβάνω η κατάσταση δεν έχει οριστικοποιηθεί. Πάντως συνάντησα ε, τον ε, Ομοσπονδιακό Υπουργό Υγείας της Γερμανίας. Ε, συζητήσαμε για μία ώρα και ένα τέταρτο με απόλυτη ειλικρίνεια και νομίζω ότι ο Γερμανός υπουργό άκουσε αυτά που του είπα. Ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν μπορεί να γίνει με μια εναρμόνιση προς τα κάτω, αλλά μια σταδιακή εναρμόνιση προς τα πάνω. Για τους νοσοκόμους, τις νοσοκόμες, ε, η κατάλληλη γραμμή είναι η 12 κάτι που είναι ε, βήμα πρόοδου βέβαια και για τη Γερμανία και για άλλες χώρες που έχουν δεκαετές πρόγραμμα σπουδών, συνεχίζονται οι συζητήσεις για να δούμε κατά πόσο οι χώρες αυτές θα μπορέσουν να συνεχίσουν για μια μεταβατική περίοδο αυτή τη δεκαετία, το δεκαετές πρόγραμμα εργασιών, υπό τον όρο όμως ότι θα αναθεωρήσουν, θα παρεξετάσουν ένα κατάλογο δεξιοτήτων για, τα, για το επάγγελμα των νοσηλευτριών και μάλιστα ο κατάλογος αυτός των δεξιοτήτων θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά γιατί είναι ραγδαίες εξέλιξη το επάγγελμα του νοσηλευτή. Δεν μπορούμε λοιπόν ε, να, διακινδυνεύουμε εδώ την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών. Επαναλαμβάνω, η συζήτηση είναι ανοιχτή. Δεν υπάρχει αδιέξοδο μεταξύ μας. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα με το Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μάλιστα είναι πιο προηγμένο σε σχέση με το Συμβούλιο στη συζήτηση για τις νοσηλεύτριες. Ελπίζω πάντως ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία, αν και προς το παρόν δεν το έχουμε καταφέρει. Και πιστεύω ότι θα είναι ακαθόδηση συζήτηση. Αυτά προς το παρόν αγαπητοί συνάδελφοι. Το θέμα αυτό με προβληματίζει μέρα και νύχτα ολόκληρες εβδομάδες. Προχωρούμε αργά αλλά σταθερά. Έχουμε αρκετές δυσκολίες και αν βρούμε λύση θα είναι ένα πολύ χαρμόσυνο μαντάτο και μια πολύ καλή αρχή για το 2013. Και ευχαριστώ και τους βουλευτές και τους βοηθούς τους που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Ένα μείζωνο σημασία θέμα για τους ε, συμπολίτε μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση της πρόοδου που έχει σημειωθεί και της πρόοδου που πρέπει ακόμα να σημειωθεί. Σας ευχαριστώ για το ότι Προσπαθείτε συνεχώς να επιτύχετε συμφωνία, αρκά ή γρήγορα θα πρέπει να ψηφίσουμε. Βεβαίω, δεν μπορεί να συμφωνούμε όλοι σε όλα, αλλά ξέρω ότι κάνετε κάθε προσπάθεια. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε τις απόψει των σχεδόν συγγενών, ξεκινώντα με την Constance Λικρύπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχηθώ ότι καλύτερο στα μέλη της Επιτροπής Θέλω προσωπικά σε όλους να ευχηθώ ένα εξαιρετικό νέο έτος 2013. Για το θέμα της αναγνώρισης λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι ένα θέμα στο οποίο θα συνεχίσουμε από ό,τι φαίνεται κάποιες συζητήσεις αναζητώντας ε, ορισμένες συμβιβαστικές ε, λύσεις στα πλαίσια του πνεύματος συνεργασίας. Υπάρχουν διαφορές ε, και μάλιστα όχι μόνο σε λεπτομέρειες αλλά και σε πιο σημαντικά θέματα στα οποία θα πρέπει να εμβαθύνουμε. Η συγγήτρια είπε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια, να προσπαθήσουμε να εξομαλύνουμε κάπως τις διαφορές και να καταλήξουμε σε μια ισχυρή πλειοψηφία έτσι ώστε η συμμετοχή μας στις διαπραγματεύσεις ε, να είναι συνεκτική και αποτελεσματική. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Κάρτα νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει για το θέμα των προθεσμιών εδώ. Ε, πρέπει να συζητήσουμε το θέμα και με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με το εφικτό της διαδικασίας για τη σιωπηλή αδειοδότηση. Όπως είπε και η συγγήτρια, θα πρέπει να σεβαστούμε τη συγκεκριμένη αυτή αρχή. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό μέσο διαπραγμάτευσης με τα κράτη-μέλη και έτσι θα μπορέσουμε να τα υποχρεώσουμε να προχωρήσουν στην έκδοση αυτής της Ευρωπαϊκής Κάρτας. Ακούμε βέβαια τις ανησυχίες ορισμένων χωρών και τις ανησυχίες των εργαζομένων στον κλάδο της υγείας. Και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να συμφωνήσουμε πάνω σε μια προθεσμία προσωρινής διακοπής έτσι ώστε να υπάρξει η σωστή ενημέρωση από πλευράς των ενδιαφερομένων. Η έμεση αυτή αδειοδότηση δεν στοιχειοθετεί αυτόματο δικαίωμα άσκησης ιατρικού, η συγκεκριμένη περίπτωση επαγγέλματος. Στα υπόλοιπα θέματα νομίζω ότι είμαι ικανοποιημένη από την πρόοδο που έχει σημειωθεί και λαμβάνουμε υπόψη οι συζητήσεις της θέσης μας. Οι τροπολογίες που έχουν γίνει δεκτές θα πρέπει να είναι σωστά πλαισιωμένες, να εξετάζονται κατά περίπτωση σχετικά με τη μερική πρόσβαση πάντα. Και αυτό δεν αφορά φυσικά τα επαγγέλματα στα οποία υπάρχει ήδη άμεση αναγνώριση των επαγγελματικών ικανοτήτων. Λάβαμε υπόψη τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει ορισμένες επαγγελματικές κατηγορίες και γι' αυτό οι τροπολογίες μου για λόγους γενικού συμφέροντος, σαν παράδειγμα, είναι θέματα που θα πρέπει να περνούν και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και συμπεριλαμβάνεται η πρόταση αυτή στις συμβιβαστικές τροπολογίες. Για αυτούς τους λόγους διευκρινίζουμε ότι ένα κράτη μέλος θα μπορεί να απορρίψει ε, μια αίτηση μερικής πρόσβασης και αυτό είναι κάτι το οποίο θα καθησυχάσει θα έλεγα πολλούς από τους εμπλεκόμενους στη συζήτηση. Να διευκρινίσω ότι αυτή η βασική αρχή η οποία προέρχεται από την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα πρέπει να γίνεται σεβαστή. Σε μια τροπολογία μου υπογραμμίζω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν οδηγούνται στην απόρριψη μιας αίτησης μερικής πρόσβασης. Κατανοώ ότι μια τέτοια διαδικασία δεν είναι πάρα πολύ σε εισαγωγικά χρηστική, βολική και δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάζει σε ημερήσια βάση ε, κάποιες αιτήσει. περιπτώσει απόρριψη δηλαδή αίτηση μερική πρό, ε, πρόσβασης. Παρ' όλα αυτά, εδώ θα πρέπει ε, να ε, εφαρμόζεται το άρθρο 60 σχετικά με τον απολογισμό αναδιετία και σχετικά με τη δυνατότητα να συμπεριληφθεί η μερική πρόσβαση στην διετή αυτή, αναδιετία μάλλον, αξιολόγηση για τα στάζ. Είδα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της οδηγίας της και κάνει εδώ μια θαραλέα πρόταση, εντάσσει τα στάζω στα πλαίσια της οδηγίας, εγώ θα ήθελα να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο έτσι ώστε να υπάρξει ένα ποιοτικό πλαίσιο για τα στάζου και στα πλαίσια μιας αιτιολογικής σκέψης αλλά και στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου άρθρου. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την πρωτοβουλία αυτή για να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα για την σημασία της ποιότητας της διαδικασίας των στάζων. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε την διαπραγμάτευση έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια σωστή βάση συζήτησης με το Συμβούλιο και τα άλλα όργανα. Επιμένω λοιπόν στο συγκεκριμένο θέμα πλαισίωση σωστή της διαδικασίας αναγνώρισης των στάζ. Μια τροπολογία, η 639 Σφάμπ και Κάρας αφορούν το 55α μικρό λέει ότι ένα στάζ δεν θα πρέπει να υποκαθιστά την σωστή εξέταση ε, από την οποία θα πρέπει να περνά ένας υποψήφιος για να ενταχθεί σε μια επαγγελματική κατηγορία ανάλογα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν στην χώρα προέλευσης. Νομίζω ότι και εδώ θα καταλήξουμε σε μια κάποια συμφωνία εύκολα. Τελειώνοντας, όπως και η συγγήτρια, θα αναφερθώ σε δύο ε, επαγγέλματα απόλυτα σεβαστά που εκφράζουν πολλά επιχειρήματα και επάνω στα οποία θα έλεγα έχουμε ήδη αφιερώσει αρκετό χρόνο και ενέργεια. Τους συμβολεογράφους και τους νοσοκόμους νοσοκόμες. Για τους συμβολιογράφους σας είμαστε ειλικρινεί. Εδώ υπάρχει μια διέρεση ανάμεσά μας και στη δική μας επιτροπή και στα άλλα όργανα. Ακούμε διαφορετικές απόψεις, ακούμε επιχειρήματα που καταθέτουν οι εκπρόσωποι της ε, κατηγορίας αυτής που είναι πολύ διστακτική για την ένταξή του στην οδηγία. Νομίζω ότι και στο Συμβούλιο τα πράγματα παρουσιάζονται ιδιαίτερως περίπλοκα και η συμπερίληψη της επαγγελματικής κατηγορίας αυτή στην οδηγία τίθεται θα έλεγα με τρόπο οξύτατο. Καταρχήν υπάρχουν αυτοί που προωθούν την ασφάλεια, θα έλεγα την νομική, για την δραστηριότητα τη συμβολιογραφική. Από την άλλη θα πρέπει να, να γνωρίσουμε ότι το θέμα αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα στο Συμβούλιο, να μπλοκάρει τις συζητήσεις και να προκαλέσει καθυστερήσεις στο σύνολο της διαδικασίας υιοθέτηση αυτής της πολύ σημαντικής οδηγίας. Γνωρίζουμε ότι πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι ε, είναι ανυπόμονοι έτσι ώστε να μπορέσουν να ωφεληθούν από την οδηγία αυτή και θέλουν η διαδικασία να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν. Είχα κάνει, υπενθυμίζω, μια πρόταση πρόσφατα επί του θέματος των συμβολιογράφων ίσως θα μπορέσουμε να βάλουμε μια χρονική προθεσμία πολύ συγκεκριμένη για το επάγγελμα αυτό με πολύ ξεκάθαρο τρόπο να υπάρξει μια ρήτρα συνάντησης, μια ρήτρα λοιπόν ειδικά για τους συμβολιογράφους. Τώρα για τους νοσοκόμους, άνδρες και γυναίκες. Και εδώ θα πρέπει να βρούμε μια συμβιβαστική λύση Επί μακρόν είχαμε την δυνατότητα να εκθέσω σε προηγούμενες συναντήσεις τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Καταθέσαμε και μια τροπολογία στο άρθρο 31. Λέμε ε, ότι μπορεί να υπάρξει, συμφωνούμε σε μια βάση συζήτησης και να καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική λογική θέση. Άκουσα προσεκτικά εδώ την εισηγήτρια Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τα ειδικά χαρακτηριστικά των συστημάτων κατάρτισης που ισχύουν στα διάφορα κράτη-μέλη και θα πρέπει επίσης να καταστήσουμε πιο αναλυτική ίσως και πιο απαιτητική την λίστα αυτή των κατάλογο απαιτήσεων και να μην βασιζόμεθα αποκλειστικά στην ε, προϋπηρεσία, στα έτη προϋπηρεσίας. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να γίνουν στη συγκεκριμένη περίπτωση κάποιες επιπλέον προσπάθειες ε, εφάνταστες, δημιουργικές για να καταλήξουμε κάπου. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την δυνατότητα ύπαρξης διαφορετικών συστημάτων κατάρτισης χώρα που είναι σημαντικά για ορισμένες χώρες. Τελειώνοντας με μία φράση, εργαστήκαμε πολύ βλέποντας τις διάφορες διεκδικήσεις που υπάρχουν τις ανησυχίες και τις συνεισφορές των διαφόρων τομεακών κατηγοριών. Έχει κάνει σημαντικά βήματα η συγγήτρια και γι' αυτό θα πρέπει να καταλήξουμε πλέον σε ένα οριζόντιο όραμα και να μπορέσουμε έτσι να συνθέσουμε μια τελική θέση η οποία να είναι προϊόν συνεκτικής σύνθεσης όλων των βημάτων στα οποία έχουμε προχωρήσει στον τομέα της εναρμόνισης ε, στους διάφορους τομείς. Πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε ένα οριζόντιο σφαιρικό ε, όραμα, σε μια σφαιρική αντίληψη. Ε, θέλουμε την κινητικότητα, θα φέρει ανάπτυξη και θα δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ενδιαφέροντα σχόλιά σας σε αυτά τα οποία είπε η κυρία Βρίνιο. Η κυρία Τούρινεν επίσης πρέπει να πάει και στην Επιτροπή Οικονομικών. Ε, αν δεν πειράζει την κυρία Παρβάνοβα θα ήθελα να ακούσουμε πρώτα την κυρία Τούρινεν και μετά τις κυρίες ε, Παρβάνοβα και Μακλάρκιν. Ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά σε όλους ε, και στην εισηγήτρια. Έχουμε λίγες αλλά σημαντικές ανησυχίες. Νομίζω πως πλησιάζουμε σε κάποιο τέλος. Επίσης θεωρώ πως θα μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου την επόμενη εβδομάδα, αλλά θα χρειαστεί σκληρή δουλειά. Και θέλω να αναφέρω τις ανησυχίες που έχουμε ακόμα. Πρώτα απ' όλα για την μερική πρόσβαση. Είδα την διατύπωση και ανησυχούμε για το τελευταίο κομμάτι του άρθρου 4 το Συμβούλιο το διέγραψε και νομίζω πως το ίδιο πρέπει να κάνει και το Κοινοβούλιο για την πρακτική άσκηση. Το ζήτημα είναι λοιπόν το αν μπορεί να διαχωριστεί η δραστηριότητα και αν ορίζεται από το καθεστώς του επαγγελματός ως αυτόνομο επάγγελμα στο ε, κράτος υποδοχής ή προέλευσης. Εμείς θέλουμε να σβήσουμε το κομμάτι του κράτους προέλευσης. Για την πρακτική ασκή, όσο και αν ε, αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε για να υπάρχουν ποιοτικές ε, πρακτικές ασκήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, ήταν αυτό και στην έκθεσή μου του 2010, είναι κάτι που μας ανισχύει, το στηρίζω, αλλά όπως ανέφερα, στις 5 Δεκεμβρίου η Κομισιόν ξεκίνησε τη διαβούλευση της δεύτερης φάσης ακριβώς για αυτό το ζήτημα με τους κοινωνικούς εταίρους και ίσως είναι κάπως πρόωρο να ξεκινήσουμε να ρυθμίσουμε το ζήτημα σε επίπεδο σύμβασης σε αυτή την οδηγία. Δεν ξέρω αν είναι η σωστή στιγμή και το σωστό σημείο να γίνει αυτό. Αλλά είδα την πρόσφατη πρότασή σας που είναι πολύ περιορισμένη και ίσως αποτελέσει μια λύση. Γιατί βέβαια πρέπει να δουν και οι κοινωνικοί εταίροι το τι μπορεί να γίνει. Για τις γλώσσες, όπως ξέρετε, ξέρετε πως εμείς είμαστε οι πράσινοι και Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία ε, και έχουμε μεγάλη ευαισθησία για τις γλώσσες και καμιά φορά ίσως χρειάζονται δύο γλώσσες εδώ πέρα λέει μία από τις επίσημες ε, θα το ξαναδώ έτσι ώστε όλη μου η ομάδα να είναι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα αυτό. Το σημείο 4. Πράξεις κατεξουσιοδότηση. Νομίζω πως Πρέπει και αυτό να το δούμε βάθος και να βρεθεί μια λύση ειδικά όσον αφορά το κοινό πλαίσιο εκπαίδευση γιατί είναι πολύ ευαίσθητο ζήτημα αφορά τη διδακτέα ύλη, τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα και θέλουμε να διασφαλίσουμε πως η αρμοδιότητα λήψη αποφάσεων θα βρίσκεται στα επαγγέλματα τα ίδια. Επίσης, εύκολα. Νομίζω μπορούμε να ζητήσουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Είναι καλό να συναντιόνται επαγγελματικέ ενώσει, αλλά ε, είναι κάτι που πρέπει να ξεκινήσουν οι ίδιες. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις νοσοκόμες και τους νοσηλευτές. Θέλουμε πως θέμε μια ρεαλιστική λύση. Η Χάιντι είναι από τη Γερμανία, έχουν το διπλό σύστημα, είναι η συντονίστριά μου. Και εμεί στη Δανία έχουμε το διπλό σύστημα, ξέρω λοιπόν τι είναι. Έμαθα επίσης πως υπάρχουν διαφορετικές δομές στα νοσοκομεία. Στη Δανία έχουμε νοσηλευτές και βοηθούς νοσηλευτές. Δεν το έχουν αυτό στη Γερμανία. Υπάρχουν μόνο νοσηλευτέ και βοηθοί ιατρού. Διαφορετικέ δομέ. Αν θα μπορούσαμε λοιπόν να σεβαστούμε τις διαφορές, ε, αλλά να έχουμε ακόμα συνθήκες υψηλής ποιότητας, νομίζω πως θα είναι κάτι καλό. Μία λύση θα ήταν να δούμε τι, κάναμε, τι κάνατε για τους γιατρούς και άλλη μία δεν ξέρω αναφέρατε ε, κάπου που κοιτάτε περισσότερο το περιεχόμενο μπορούμε να δούμε νομίζω μια λύση, δεν ξέρω αν θα είναι τα 10 ή τα 12 χρόνια που θα καθορίσουν την ποιότητα ε, ενό νοσηλευτή. Ε, σα ευχαριστώ λοιπόν και για την ευελιξία που δείξατε. Πάω τώρα στην Επιτροπή Οικονομικών και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Ωραία, σα ευχαριστώ που εστιάζετε στα ζητήματα όπου πρέπει να σημειωθεί πρόοδος. Η κυρία Παρβανόβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχηθώ καλή χρονιά σε ολόκληρη την Επιτροπή. Επίση ζητώ συγγνώμη ο κύριο, εξ κύριου Κριστιαν Μπουσόη ο οποίο δυστυχώ ουσιάζει. ευχαριστή την συγκεκριά και τις κοιόδε συγκεκρίες για τη στενή συνεργασία σε γενικέ γραμμέ, ο συναδελφό μου είναι υπέρ των συμβαστικών προτάσεων και ελπίζει και τα υπόλοιπα ζητήματα να λυθούν τι επόμενε μέρε, ε, για να ανοίξει έτσι ο δρόμο για μια ευρεία συμφωνία στην Επιτροπή μα. Τώρα θα διατρέξω τα σχόλιά του. Πρώτα απ' όλα για την μερική πρόσβαση. Πρέπει να φροντίσουμε η μερική πρόσβαση να παραμείνει κάτι που θα είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Γι' αυτό στηρίζουμε πλήρως την συμβαστική πρόταση καθώς δεν θα καλύπτονται έτσι τα επαγγέλματα που έχουν αυτόματη ε, αναγνώριση και βεβαίως θα υπάρχει δυνατότητα να αρνηθούμε αυτή την πρόσβαση για γενικούς λόγους ε, δημοσίου συμφέροντος όπως ορίζει το, 10. το Τέλος ε, για την πρακτική άσκηση ειδικά όταν είναι προαπαιτούμενο για κάποια επαγγέλματα είναι κάτι το σημαντικό για την ε, ε, πρόσβαση και βέβαια πρέπει να γνωρίζονται όλες οι πρακτικές ασκήσεις και όχι μόνο οι αμοιβόμενε. Υπάρχει όμως ε, μια πτυχή στο άρθρο 55α που πρέπει να δούμε. Η διάταξη για την αναγκαιότητα πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο μια σύμβαση που θα ορίζει τουλάχιστον τους μαθησιακούς στόχους ίσως παρά είναι περιοριστική. Οι συμβάσεις δεν περιέχουν ε, όλες αυτές τις πληροφορίες και δεν πρέπει να επιβάλλουμε τέτοιο βάρος εάν δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Για τις προθεσμίες, για την ε, σιωπηλή εξοδότηση. Θεωρούμε πως θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προθεσμίες για να λειτουργήσει κάτι τέτοιο, οπότε καλό είναι το κράτος προέλευση να έχει τρεις εβδομάδε για τη δημιουργία επαγγελματική κάρτας και να έχουμε διατάξεις για την άρση των διατάξεων αυτών εάν ζητηθούν περισσότερες πληροφορίες από το κράτος προέλευσης, ειδικά όταν έχουμε συνέπειες για την ασφάλεια των ασθενών. Για το μηχανισμό ειδοποίησης πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο σύστημα και θεωρούμε πω η δημιουργία ενό μηχανισμού ε, ειδοποιήσεις θα συνεισφέρει αυτό, αλλά πρέπει βεβαίως να δούμε το πώς θα σημαίνει ο συναγερμός και βεβαίως δεν θα πρέπει να σημαίνει ο συναγερμός πριν ληφθεί η οριστική απόφαση από κάποιον αρμόδιο φορέα, είτε είναι κάποιο πειθαρχικό είτε κάποιο δικαστήριο στην ε, χώρα υποδοχής και βεβαίως θα πρέπει πάντα να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο αθωότητας και να μην ε, ξεκινάει κάποια έρευνα εφόσον δεν τίθεται να αμφιβόλω η επαγγελματική επάρκεια. Τώρα για τις, ε, τις γλωσσικές εξετάσεις έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, η τροπολογία 605 τώρα καλύπτει νομίζω τα στοιχεία που πιστοποιούν τη γνώση γλώσσας δεν πρέπει πάντα να γίνονται εξετάσεις από τις αρμόδιες αρχές απευθείας πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα να χωρίσουν αρμοδιότητα αυτή ε, επίσης ε, θα είναι ίσως καλύτερο να γίνεται υπό να γράψουμε τη λέξη υπό την εποπτεία αντί για υπό την ευθύνη γιατί αυτό δεν είναι κατά κατά κύριο λόγο αρμοδιότητα των αρμοδίων αρχών και μπορούμε νομίζω να προσαρμόσουμε αναλόγως ε, και τη διατύπωση του, της αιτιολογικής σκέψης. Για την βασική εκπαίδευση των ιατρών τώρα υπάρχει μια απέτηση η οποία λέει πως θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 ε, έτη και 5.500 ώρες ε, πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης. Η συμβαστική λύση που προτείνει ο εισηγητής για 6 χρόνια και 5.500 ώρες είναι ένας κανόνας και η δυνατότητα βεβαίως υπάρχει να διατηρηθούν πενταετή προγράμματα αρκεί να γίνονται σεβαστά, σεβαστές προδιαγραφές της οδηγίας για να βγούμε από αυτή τη δυσκολία. Εν πάση περιπτώσει, όπως έγινε και για άλλα επαγγέλματα, η περίοδος ε, εκπαίδευσης σύμφωνα με τις μονάδες ECTS ε, δεν θα πρέπει να εκφράζεται μόνο σε τέτοιες μονάδες καθώς δεν είναι ομοιόμορφη ε, η βαθμολόγησή τους. Και τέλος πρέπει να δούμε πως έχουμε και το ζήτημα της αξιολόγησης ε, των νοσηλευτών. Σας ευχαριστώ και πράγματι για αυτό το οποίο είπατε είναι κάτι στο οποίο αναμένουμε λύση από την κυρία Βανιό. Η κυρία Μακλάρκιν, α, και υπάρχει και ο κύριος η κυρία Χάνσλικ ε, και άλλοι στον κατάλογο μιλητών. Αν θέλει και άλλος λοιπόν να μιλήσει, να, να πει κάτι, μπορεί να μου κάνουν νόημα. Κυρία Μακλάρκιν. Ευχαριστώ και καλή σας χρονιά. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ και σας προσωπικά πρόεδρε για το βραβείο και το, ε, την αναγνώριση σας ε, στην ε, οικονομία Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν για αυτή τη διάκριση. Σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Φυσικά τώρα αρχίζει η καινούργια χρονιά, αλλά θέλουμε να επιλύσουμε τα ακριβή προβλήματα του 2012. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες ε, και πρόοδο σε τεχνικό επίπεδο. Θα επικεντρωθώ σε ορισμένα μόνο θέματα που είναι σημαντικά για τους συντηρητικούς μεταρρυθμιστές για τις συμβαστικές λύσεις και κυρίως για τη βασική ιατρική εκπαίδευση. Αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. δεν είμαστε ικανοποιημένοι ακόμη από τη συμβαστική λύση, γιατί προβλή, προβλέπεται παρέκκληση σε έκτακτες περιστάσεις. Αυτό δεν μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, γιατί έχουμε υψηλές προδιαγραφές στο Ηνωμένο Βασίλειο και αν υψηλή ιατρική εκπαίδευση μπορεί να εξασφαλιστεί σε 5 χρόνια και 5.500 ώρες, γιατί να αναγκαστούν τα πανεπιστήμια να παρατείνουν τον κύκλο σπουδών. Δεν έχει νόημα αυτή η πρόταση και αν ε, δώσει καλύτερα πιο βάσιμα επιχειρήματα η κυρία Βερνιά για την πρόταση, ε, να τα συζητήσω, αλλά ούτε καν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με αυτό. Επίση, για τα τομεακά επαγγέλματα με ανησυχούν οι τροπολογίε, γιατί επαφείται στα κράτη-μέλη να οργανώσουν ε, τα εκπαιδευτικά του συστήματα. Και φοβάμαι ότι θα παρεύουμε σε συστήματα που ισχύουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και λειτουργούν πολύ καλά. Δεν θέλουμε μία ενιαία προσέγγιση για όλου, ε, ανεξάρτητα των ιδιαιτερότητων. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό ο στόχο τη οδηγία. ό,τι αφορά τη συμβεστική λύση για τι ε, πρακτικέ ασκήσεις. Η οδηγία αυτή δεν αφορά την εργασία και τα κοινωνικά δικαιώματα, αλλά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Και γνωρίζετε τη ε, γνώμη μας για το 50α, που μιλά για, τα, ε, για τους ε, εκπαιδευτικούς στόχους της πρακτικής άσκησης. Δεν νομίζω ότι είναι εντός θέματος αυτή, αυτό το άρθρο. Επαναλαμβάνω, μιλούμε για τα επαγγελματικά προσόντα σε ό,τι αφορά τα κοινά πλαίσια εκπαίδευσης και κατάρτισης. Προτείνει η να ισχύσουν και για τους γιατρούς, νοσηλευτές και τις ΜΕΣ και ΜΕΦΤΗΡΕΣ. Δημιουργείται ένα επιπλέον, μια επιπλέον περιπλοκή στην αναγνώριση, ε, κάτι που βαίνει βάρος και των αρμοδίων αρχών και των επαγγελματιών. Εμείς θέλουμε να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες. Αυτός είναι ο στόχος έκθεσης και ε, όχι να είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι και να προσπαθήσουμε να τρέξουμε πριν καν να αρχίσουμε να περπατάμε. Σε ό,τι αφορά τις γλωσσικές εξετάσεις, ε, να μιλούμε για υποπτία ή έλεγχο και όχι ευθύνη. όπως προβλέπουν κάποιες τροπολογίες. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν είναι όλες οι αρμόδιες αρχές ε, αυτές που έχουν την ευθύνη της ε, διοργάνωση αυτών των γλωσσικών ε, εξετάσεων, αρκεί η εποπτεία ή ο έλεγχός τους. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη της συγκήτριας. Επίσης, ε, αυτό που λέμε πριν την πρόσβαση για το επάγγελμα, να ξέρουμε ότι θα προηγούνται οι γλωσσικές αυτές εξετάσεις πριν την πρόσβαση στο επάγγελμα. Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική ταυτότητα, καλή πρόταση. Βέβαια, προτείνονται κάποιες διορίες μόνο για τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης και όχι της χώρας υποδοχής. Και όμως η χώρα υποδοχής είναι αυτή που θα αναγνωρίσει τα επαγγελματικά προσόντα. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να επανεξετάσουμε και αυτό το θέμα. Γιατί πολλές τροπολογίες επισήμαναν αυτή την ανησυχία. Πάντως αυτά είναι τα χέρια για μας θέματα. Έχω παραλείψει ε, με ιδιαίτερη επιτυχία το θέμα των νοσηλευτριών, πάντως προσβλέπω σε ανέβρεση επικοδομητικών λύσεων για τα επαγγέλματα αυτά. Και θα έχουμε πιστεύω κάποια φορά συνεργασία με τους κοιόδης συγκεκριτές και την συγκεκριτές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ λοιπόν που εκφραστήκατε σε όλα αυτά τα θέματα. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να εντοπίσουμε σωστά τα σημεία στα οποία πρέπει να υπάρξει μια συμβιβαστική λύση. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Δεν θέλω να εμποδίσω τη συζήτηση, αλλά να ενθαρρύνω τους υπόλοιπους ομιλητές να είναι σύντομοι. Ο κ. Σφάμπ δεν είναι εδώ. Έχει εγγραφεί, αλλά δεν τον βλέπω. Χάσλεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχηθώ θερμά ευτυχές στο νέο έτος. Θα είμαι εξαιρετικά λακωνική. Κυρίως θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την εισηγήτρια για το πολύ αξιόλογο έργο της, παρόλο που ήταν περίπλοκο και εξαιρετικά δύσκολο. Και θα ήθελα να σχολιάσω κάποιες συμβαστικές τροπολογίες. Ό,τι αφορά τη μερική πρόσβαση στο σημείο 4 του προημίου και στο άρθρο 4F προτιμώ για το θέμα της υγείας να το αναφέρουμε και ε, το θέμα της αυτόματης αναγνώρισης για κάποια επαγγέλματα και το θέμα των κοινών πλαισίων εκπαίδευση και των εξετάσεων. Σε ορισμένε περιπτώσει, τομεακά επαγγέλματα μπορούν να αναγνωρίζονται στο γενικό σύστημα. Αυτό είναι η μόνη παρατήρηση που έχω για τη μερική πρόσβαση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες, ε, το άρθρο 4C και 4D αναφέρεται οι δύο εβδομάδες και μία εβδομάδα. Στο 56, στο 56 έχουμε 48 ώρες θεωρώ ότι είναι κάπως ε, σύντομες αυτές οι προθεσμίες. Γιατί σε τελική ανάλυση θέλουμε να επισπεύσουμε αυτή τη διαδικασία, αλλά θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές στις προθεσμίες μας και να είναι εύκολη η τήρησή τους. Δεν είμαι βέβαιη ότι οι προθεσμίες που προτείνουμε είναι οι πιο λογικές. Θα μπορούσαμε να το αναθεωρήσουμε αυτό το θέμα. Και ένα άλλο θέμα, δεν ξέρω αν επιδέχεται περαιτέρω διαπραγμάτευση, θα μας το πει η συγγήτρια, με προβληματίζει ο μεγάλος αριθμός ορών που απαιτείται στο άρθρο 41 για τις ε, ΜΕΕΣ, 5.000 ώρες, γιατί στην ε, Πολωνία έχουμε 4.700 ε, ώρες και κάτι. Δεν φτάνουμε στις 5.000 ώρες. Δεν ξέρω αν επιδέχεται να περαιτέρω αυτό το θέμα, αλλά θα ήθελα να σε επισημάνω αυτό το πρόβλημα που έχουμε στην Πολωνία για την βασική εκπαίδευση των μεών και μευτήρων. Επίσης, το θέμα των νοσηλευτιών των Πολωνο, της Πολωνίας, άρθρο 33 και το θέμα των μεών στην Πολωνία. Το θέμα αυτό προβληματίζει όχι μόνο Πολωνούς αλλά και άλλους συναδέλφους και έχουν κατατεθεί τροπολογίες όχι μόνο από Πολωνούς νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μία λύση για τις πολωνέζες ε, νοσοκόμες, γιατί νομίζω ότι πολλοί περισσότεροι βουλευτές έχουν πια συμφωνήσει για τη διευθέτηση αυτού του θέματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτά. Ευχαριστώ ε, κύριε Βερχαήλ. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ και την κυρία Βασκέμπε, η οποία βεβαίω έχει συνεργαστεί με την εισηγήτρια για αυτά τα θέματα το ερώτημά μου το αναφέρατε κυρία Ρεβενιού όπως μιλήσατε και με τον κύριο Μπα, τον αρμόδιο Γερμανό Υπουργό. Το ζήτημα όμως είναι πώς βλέπετε και τις ε, τροπολογίες ε, των επιτροπών για, τις, για τους ε, νοσηλευτές και το διπλό σύστημα που υπάρχει στη Γερμανία καθώς υπάρχουν πολλές ώρες θεωρίας με την παράλληλη πρακτική εκπαίδευση. Πώς βλέπετε λοιπόν τις ε, τροπολογίες ε, από την Επιτροπή. Γιατί η υπουργική πλευρά είναι ζήτημα του Συμβουλίου. Αλλά πρέπει να συζητήσουμε νομίζω και την θέση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστώ. Είμαι σίγουρος πως η κυρία Βερνιό θα τα απαντήσει. Δεν υπάρχουν άλλοι βουλευτές που θέλουν το λόγο. Θα ζητήσω λοιπόν τον κύριο Γιώργεν Τίτσερ να πει κάποια λόγια και μετά θα δώσω τον λόγο στην κυρία Βερνιό. Γιώργεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Θα είμαι σύντομος, αλλά θα σας εκφράσω και τις ευχές μου. Θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τις συμβιβαστικές τοπολογίες. Καταρχάς, για την Ευρωπαϊκή Κάρτα υποστηρίζουμε πλήρως τις προτάσεις σας. Παρακολουθήσαμε εμείς και τη συζήτηση για τα στάζ, τα αμοιβόμενα. Νομίζω ότι ε, μπορούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση να αλλάξουμε τη δική μας θέση, ίσως με κάποιες διορθώσεις, όχι μόνο να εμείνουμε στο θέμα της κατάστασης στη χώρα προέλευσης, αλλά και στη χώρα προορισμού. Ε, στο κείμενο αυτό δεν είναι κάτι το πάρα πολύ ξεκάθαρο, αλλά είναι μια ιδέα που θα την δεχτούμε. Μερικές φορές ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες και γι' αυτό θα πρέπει να περάσουμε σε επιμέρους επαγγέλματα. Τέσσερα από αυτά θα με απασχολήσουν νοσοκόμοι, νοσοκόμες. Ε, θα συνεισφέρομαι σε μία συμβιβαστική πρόταση. Θέλουμε να βρούμε μία λύση με τρεις βασικές λέξεις. Πραγματιστική, φιλόδοξη και ευρωπαϊκή. Μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό επάγγελμα. Έρχομαι τώρα στο θέμα της εφαρμογής επιβολής. κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για τον τρόπο που πρέπει να προχωρήσει, αλλά ενημερώστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους κανόνες που ισχύουν. Αν δοθούν εξαιρέσει, αποκλήσεις, όπως γίνεται για τους γιατρούς σαν παράδειγμα, το θέμα είναι ποιος θα ελέγξει και ποιος θα επιβάλλει τις αποκλήσεις αυτές, ποιος θα τις εφαρμόσει καλύτερα. και τέτοιες εξαιρέσεις αν συζητήσουμε ας πούμε θέματα διεύρυνσης στο μέλλον είναι θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τις υποψήφιες χώρες, έχουν σημασία. Πάντως θέλουμε κανόνες, αρκεί οι κανόνες αυτοί να είναι εφαρμόσιμοι και ελέγξιμοι. Άλλο επάγγελμα, αρχιτέκτες, αρχιτέκτονες. Δύο παρατηρήσεις. φαίνεται ότι η ελάχιστη περίοδος είναι μεγαλύτερη από η αδίποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο συμβαίνει κάτι τέτοιο. Συμβαίνει για τους ιατρούς, συμβαίνει για τους οδοντίατρους, γιατί συμβαίνει για τους αρχιτέκτονες. Τώρα για την Ισπανία. Πενταετής περίοδος προβλέπεται στην Ισπανία και όχι εξαετής όπως προτείνεται. Αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε. Για τους συμβολιογράφους συνειδητοποιούμε ότι το επάγγελμα αυτό δεν είναι έτοιμο να συμπεριληφθεί στην οδηγία αυτή, το εκτιμούμε έτσι. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο κομψό για να μην του συμπεριλάβουμε, λέγοντας ότι θα συνεχίσουμε τις επαφές για περαιτέρω ένταξη του επαγγέλματος αυτού στη λίστα. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος η κυρία Βερνιό θα κλείσει τη συζήτηση. Σύντομα παρακαλώ. Γιατί βλέπω ότι ο κύριος Ζουβά είναι εδώ για το επόμενο θέμα. Θα είμαι σύντομη. Δεν τα σημείωσα όλα και δεν μπορώ, δεν έχω το χρόνο να απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά. Πάντως θα πρέπει νομίζω να συνεννοηθούμε πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Λεγκρίπ για μια σφαιρική και οριζόντια αντίληψη των πραγμάτων. να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αν καταφέρουμε να είμαστε πραγματικοί και φιλόδοξοι και Ευρωπαίοι, αυτό, αυτό ακριβώς θέλουμε. Νομίζω ότι τα τρία αυτά επίθετα, οι τρεις αυτοί επιθετικοί προσδιορισμοί είναι αυτό που θέλουμε. Θαύματα εγώ δεν κάνω παρότι έχω το όνομα της Μπερναντέτ, της Λούρδης, αλλά παρόλα αυτά ανοίξαμε νομίζω κάποιες δυνατότητες και ανοίξαμε επίσης και τη δυνατότητα να απεμπλακούμε από την υπόθεση των συμβολιογράφων. Την Τετάρτη το απόγευμα θα συναντηθούμε με όλους τους σκιώδεις για τα κομβικά θέματα Είχα επίσης μια συνάντηση να πω εδώ και με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό των Γερμανών, τον κύριο Μπάρ. Η συζήτηση δεν έχει κλείσει και δυστυχώς δεν θα κλείσει εύκολα. Παρ' όλα αυτά προσπαθήσαμε ο καθένας να κάνουμε ένα βήμα προς την κοινή κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να μην μπλοκάρουμε ο καθένας σε επίπεδο εθνικού εγωισμού, θεσμικού ευρωπαϊκού εγωισμού, Ελπίζω να καταλήξουμε σύντομα σε μια λύση. Σχετικά. Ε, ε, σας έγινε και μια ερώτηση για τις ε, τροπολογίες. Ναι, πρώτα με τους σκιώδες ηγητέ. Οκ. Οπότε, να υπενθυμίσω τις ημερομηνίες. Θα ψηφίσουμε το πακέτο υπό την ίδια της κυρίας Βερνιό στις 23 Ιανουαρίου, σε δύο εβδομάδες, στην επόμενη μας συνεδρίαση, δηλαδή αμέσως μετά το Στρασβούργο. Θα είναι μια γεμάτη μέρα γιατί θα ψηφίσουμε και για τις παραχωρήσεις και το μείζον πακέτο για τις δημόσιες συμβάσεις, δημόσιες προμήθειες. Ευχαριστώ την κυρία Βερνιό, τους σκιώδη ηγητές, τον κύριο Τίτσερ εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και να σα υπενθυμίσω ότι ο κύριος Ρόρι Κουίν, ο Ιρλανδός υπουργό, ενδιαφέρεται και προσωπικά για το θέμα αυτό. Και αν δεν κάνω λάθος, ήδη έχει συναντήσει τους σκιώδη ηγητές, κάτι που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ε, και προϊονίζεται μεγάλη πρόοδο και ταχεία δεδομένης προτεραιότητας που δίνει στο θέμα αυτό η Ιρλανδική Προεδρία. Ωραία, ας περάσουμε τώρα στο επόμενο μας σημείο που προβλέπει αναθεώρηση και γενική επισκόπηση της κατάσταση του σημαντικού θέματος των παραχωρήσεων, ανάθεση βάσεων παραχώρηση και πάλι εξέταση των συμβαστικών τροπολογιών. Θα ήθελα να προσθέσω ότι τα επόμενα δύο θέματα για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ε, δεν θα είμαστε μόνοι μας, θα έχουμε και τέσσερις εμπειρογνώμονες. Θα ακούσουμε λοιπόν τις δικές τους παρεμβάσεις. Είναι πολύ χρήσιμο να μας πω τη γνώμη τους ρυθμιστικές αρχές, εκπρόσωποι ρυθμιστικών αρχών για θέματα καταναλωτών, αλλά και ε, επαγγελματίες για αυτό το θέμα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών των επενδυτικών προϊόντων. Σας προσκαλώ λοιπόν να παραμείνετε για να ακούσετε και τους καλεσμένους μας. Τώρα θα μας μιλήσει ο κύριος Ζουβά για τις ε, συμβάσεις παραχώρησης. Παρίστανται ο κύριος Παντσέρη, ο κύριος Χατζημαρκάκης εκ μέρους του κύριου Μπουσόη, κυρία Ρίλε, θα πω και εγώ δύο λόγια για την θέση της δικής μου ομάδας και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για τις συμβάσεις παραχώρησης. Ο κύριος Ζουβά, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να εξετάσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες και τις, στις συζητήσεις ε, και τις 724 τροπολογίες ε, που προσθέθηκαν στις 236 που κατέθεσα εγώ στη δική μου έκθεση φτάνουμε γύρω στις 1000 τροπολογίες για τις συμβάσεις παραχώρησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και οδησηγητές για την πολύ επικοδομητική συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Μέχρι στιγμής έχουμε αίσια διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων παρά τις ε, διαμετρικά αντίθετες απόψεις. Χάρη στην ε, ευφία όμω και τη συνεργασία θα καταλήξουμε στη συμφωνία. Είχαμε τρεις ε, συνεδριάσεις των σχεδόν εισηγητών, έξι από την δημοσίευση των τροπολογιών, η τελευταία ήταν χθε. Γι' αυτό και δεν προλάβαμε ακόμη να βάλουμε στο νηστότοπο του Κοινοβουλίου το σύνολο των συμβαστικών τροπολογιών, γιατί μερικές τι επεξεργαστήκαμε μόλις χθες. Επίσης, έμειναν ε, κάποια τεχνικά ζητήματα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω εντάχει τους ε, στόχους. Θέλουμε ένα σαφές, ε, ευανάγνωστο, ελαφρύ, αποτελεσματικό, ρεαλιστικό νομικό πλαίσιο που θα στηρίζεται σε ένα κείμενο που θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια, την αποφύγη διακριτικής μεταχείρισης, την πλαισίωση των πρακτικών, να αποφευθούν οι καταχρήσεις και ταυτόχρονα να αναγνωρίζει και να ε, εξασφαλίσει δυνατότητα ελαστικότητας και περιθώρια ε, ελιγμών και διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων αρχών στην επιλογή. Και επίσης θέλουμε την προστιθέμενη αξία ενός ευρωπαϊκού κειμένου για να ε, διελευκαθούν κάποιοι ορισμοί, να διακρίνουμε μεταξύ συμβάσεων παραχώρησης και συμβάσεων δημοσίων προμηθειών προς όφελος και των οικονομικών τελεστών και των αρμοδίων αρχών. Έχουμε αυτή τη στιγμή 114 συμβαστικέ τροπολογίε επιτάπητος. Ε, συνεχίζουμε τη συζήτηση για ορισμένε από αυτέ. Και έχουμε καταλήξει συμφωνία για αρκετά θέματα. Θα κάνω μια σύντομη επισκόπηση ακροθυγός. Σε ό,τι αφορά την αναδιαργάνωση και διευκρίνηση, αποσαφήνιση του κειμένου. Με τις συμβαστικές τροπολογίες προσπαθήσαμε να απλοποιήσουμε και να αποσαφηνίσουμε την οδηγία για να κάνουμε το κείμενο πιο ελαφρύ, πιο εύκολο, το light approach που λέμε. Έχουμε αντιγράψει πιστά κάποια σημεία των, των δημοσίων συμβάσεων. Ε, το κείμενο βέβαια είναι περίπλοκο, αλλά περίπλοκο είναι και το θέμα. Ήταν και παραμένει περίπλοκο. Χθες μάλιστα συζητήσαμε την ανάγκη να μην είναι τόσο ελαφρύ το κείμενο εξαιτία τη περιπλοκότητά του. Παρόλο παρόλο που έχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά δεν έχουμε καταλήξει σε μια τέλεια λύση, γιατί τελειότητα κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει. Κάναμε πάντως ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Δεύτερο θέμα, ορισμός ε, των συμβάσεων παραχώρησης και των συμπαρομαρτών των θεμάτων. Ε, διευκρινίσαμε του ορισμού για να γίνει διάκριση μεταξύ των δημοσίων συμβάσεων και των δια... συμβάσεων παραχώρησης, το θέμα της μεταβίβασης των κινδύνων Επίσης έγιναν διευκρινήσεις γιατί πολλές παραχωρήσεις δεν ήταν αυθεντικές παραχωρήσεις, άδειες, ε, ε, διοικητικές άδειες. Πολλά ζητήματα διαγράφηκαν γιατί δεν καλύπτονται μια και δεν συνιστούν ε, πραγματικές συμβάσεις παραχώρησης με βάση το πεδίο εφαρμογή. Διάρκεια θέλουμε περιορισμένη διάρκεια της παραχώρησης, το θέμα της απόσβεσης ε, των επενδύσεων επίσης λαμβάνεται υπόψη, το ίδιο και για τον υπολογισμό της αξίας της σύμβασης, ε, παραπροσδιορίσαμε τον ορισμό της αξίας και μάλιστα το εξομοιώσαμε και για τις συμβάσεις έργου και υπηρεσιών με βάση το τζίρο, το συσσωρευμένο τζίρο κυκλοεργασιών. Και εκεί επιδιώξαμε μία απλοποίηση αλλά και μία οικονομική λογική. Σε ό,τι αφορά τα κατόφλια. Μερικοί τάχθηκαν υπέρ κοινών κατοφλίων μεταξύ έργων και ε, υπηρεσιών. Αυτή την αρχή την εγκρίναμε και ε, ανεβάσαμε το όριο από 5 σε 8 εκατομμύρια. Βέβαια εδώ υπάρχει μια μικρή αφησημία. Σήμερα ισχύουν τα 8 εκατομμύρια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι ίσως υπάρξουν προβλήματα, όπως με τις δημόσιες συμβάσεις, σε σχέση με τις, δημόσιες μας, με τις διεθνείς συμφωνίες. Πάντως, ε, εμείς προτιμούμε ενίο κατόφλι. Σε ό,τι αφορά τον ορισμό των βασικών αρχών της οδηγίας. Καταρχήν, σημαντική πολιτική διαβεβαίωση, η διοικητική ευχέρεια των αρμοδίων αρχών. Δεύτερη αρχή, αρχή της διαφάνειας. Θα πρέπει η σύμβαση να είναι διαφανής να μην ε, διακυβεύονται φυσικά οι διατάξεις εμπιστευτικότητας. Τρίτη βασική αρχή, ε, καθορισμό, ελευθερία του, του ορισμού των ε, κοινοφελών υπηρεσιών και των συναφών υπηρεσιών. Τέταρτο, διαπραγματευτική ελευθερία των δημοσίων αρχών. Οι κρατικέ αρχέ από μόνε του καθορίζουν τη διαδικασία. Καθορίζουν του κανόνε του παιχνιδιού. Και από τη στιγμή που έχουν καθοριστεί οι κανόνε, θα πρέπει να τηρηθούν κιόλα με βάση όμως την διαπραγμάτευση. Ξαναφέραμε τη διαπραγμάτευση στο επίκεντρο της συζήτησης. Να υπάρχει ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των αρμοδίων αρχών, των αναθετουσών και των ε, διαφερομένων. Και φυσικά η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης. Για τις εξαιρέσεις, αισθενιστήκαμε ε, την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εξαιρέσεις. Προσθέσαμε κάποιες εξαιρέσεις με βάση τα αποκλειστικά δικαιώματα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και με βάσει της συνθήκες. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός αν ο νόμος προβλέπει ένα μόνο φορέα. Σε ό,τι αφορά τις ε, δικονομικές διαδικαστικές εγγυήσεις και πάλι προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θέλουμε ε, να υπάρχουν μέτρα που περιορίζουν τεχνητά την ανταγωνιστικότητα, τον ανταγωνισμό μάλλον. Το θέμα των περιβαλλοντικών προδιαγραφών Νομίζω ότι καταλήξαμε σε μια ευφυή τελικά συμβαστική λύση, προκειμένου να εξασφαλίσουμε το σεβασμό των εθνικών, κοινοτικών και διεθνών συμφωνιών για τα εργασιακά δικαιώματα, τα θέματα περιβάλλοντος και με βάση τα κριτήρια αποκλεισμού κάποιων υποψηφίων. Σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση, σε ό,τι αφορά τις ε, κοινέ μνήες, ε, σε ό,τι αφορά το κείμενο των δημοσίων ε, συμβάσεων, θελήσαμε να απλωστεύσουμε το θέμα της διακυβέρνησης και να θεσπίσουμε ένα νέο άρθρο για να μην έχουμε συστηματική παραπομπή στο κείμενο των δημοσίων συμβάσεων. Τέλος, άρθρο 11 που συζητήθηκε χθες και επιτεύχθη συμφωνία έγινε μια αναθεώρηση και διευκρίνηση του άρθρου 11 φυσικά θα πρέπει να συμπληρωθεί τελικά με ένα νέο άρθρο ή με το υπάρχουν 50 που θα αναδιατυπωθεί. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη όμως η διατύπωση. Και έτσι, χάρη σε μεταβατικές διατάξεις ε, μεγάλης διάρκειας, θα επιτρέψουμε στις αρχές που το επιθυμούν να προσαρμόσουν όχι τις δομές τους, αλλά την νομική τους οργάνωση με τη δημιουργία ενός νομικού φορέα που θα επιτρέψει τη συνέχιση κάποιων υπηρεσιών που θεωρούνται ως ποιοτικές. Τέλος, άρθρο 15, πολύ σημαντικό, για θέματα μεταξύ δημοσίου, κρατικών αρχών. Αυτό το θέμα συζητήθηκε και επ' ευκαιρία των δημοσίων συμβάσεων. Τελικά καταλήξαμε συμφωνία παρόμοια με αυτή των δημοσίων συμβάσεων. Δυστυχώς υπάρχει ακόμη μια διαφωνία που δεν έχει επιληθεί. Ε, ποιος είναι ο τζίρος που δικαιολογεί αποκλεισμό. Μερικοί θέλουν 100%, άλλοι 80%. Υπάρχει μια ψαλίδα αριθμών θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια λύση. Επαναλαμβάνω, αναμένεται οριστικοποίηση αυτών των συμβαστικών τροπολογιών. Θα ήθελα πάντως να πω ότι όταν, είχαμε δυσκο... όταν αντιμετωπίσαμε δυσκολίες με συγκεκριμένα θέματα, το πρώτο μας μέλημα ήταν να βρούμε κάποιους γενικούς κανόνες. Αλλά δεν τα καταφέραμε, γιατί ε, έτσι πολλαπλασιάζαμε τα προβλήματα και τελικά παραιτηθήκαμε από αυτή την προσέγγιση προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε στα ειδικά θέματα και να βρούμε ειδικέ λύσεις, είτε είναι αυτές μεταβατικές είτε οριστικές και όχι γενικές όπως ήταν η αρχική μας προσέγγιση. Ευχαριστώ θερμά τους και οδησηγητές για τις πολύ επικοδομητικές συνομιλίες που είχαμε, γιατί επαναλαμβάνω το κείμενο ήταν δύσκολο, περίπλοκο και υπήρχε μεγάλη διάσταση απόψεων αρχικά, αλλά καταλήξαμε τελικά σε συμφωνίες συμβαστικές για πάρα πολλά θέματα. Ευχαριστώ θερμά και τα γραμματεία μας που με βοήθησε σημαντικά, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να μην συμφωνούσαμε πάντα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά συμφωνήσαμε για μια νυφάλια ανάλυση της κατάστασης και αναζήτηση λύσης. Ευχαριστώ και τον κύριο Ταραμπέλα, γιατί παρόλο που δεν ασχολήθηκε με το θέμα των συμβάσεων παραχώρησης, μας βοήθησε πολύ το έργο του για τις δημόσιες συμβάσεις, τις δημόσιες προμήθειες. Και εμπνεύστηκα από το κείμενο αυτό, γιατί σημαντικό είναι να σταματήσει αυτή η ανομοιομορφία των διαδικασιών που οδηγεί σε μια διαφάνεια και σε διακριτική μεταχείριση. Έχουμε διανύσει πολύ μεγάλο δρόμο και μετά από ένα χρόνο συζητήσεων εξαντλητικών και διεξοδική ανάλυση καταλήξαμε σε ένα αρκετά ενδιαφέρον πιστεύω αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύμφωνα μαζί σα που σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο στο θέμα αυτό και σα ευχαριστώ γι' αυτό. Καλώς ορίζω και τον Μάρκ Ταραμπέλα που ήρθε σήμερα uh, και χτες βεβαίω είχαν κάποιε. Uh, συναντήσεις για τον δεύτερο γύρο για την οδηγία κοινοφιλών υπηρεσιών. Επίσης πρέπει να αναφέρω και την κυρία Σισκόφσκα που εκπροσωπεί εδώ πέρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρακολουθεί στενά το θέμα και ελπίζω να την ακούσουμε και εκείνη. Λοιπόν, ας ακούσουμε τώρα τους κοιόδης συγητές για τις συμβάσεις παραχώρησης. Ο κύριος Παντσέρη πρώτος. Grazie Presidente, sarò breve. Ehm, intanto vorrei anch'io ringraziare και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Ζουβά, για τις προσπάθειες που έκανα μέχρι τώρα. Θα ήθελα κάποια πράγματα να επαναλάβω. Πρώτον, έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει συμφωνία πάνω στην πρόταση. Γιατί το θέμα αυτό μαζί με τις δημόσιες προμήθειες είναι ένας τομέας καθοριστικός για την οικονομία των κρατών μελών και ιδιαίτερα των τοπικών αρχών. Οι συμβιβαστικές προτάσεις είναι καρπός μιας μεγάλης προσπάθειας, η οποία εξελίχθηκε τους προηγούμενους μήνες και καθιστούν, θα έλεγα, συγκεκριμένες τις απόψεις, ε, απλουστεύοντας ε, εν πολύ στο αρχικό κείμενο. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θα ήθελα σε κάποια σημεία να σταθώ. Πρώτον, πεδίο εφαρμογής, άρθρο 1. Εδώ έχει υπάρξει τροποποίηση. Από τη μία προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε εμείς την βασική αρχή της διοικητικής αυτονομίας και από την άλλη θα πρέπει να υπογραμμίσουμε, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να καταλάβουν μάλλον, την βασική αρχή της ελευθερίας καθορισμού της φύσης ε, των υπηρεσιών της λεγόμενης κοινή ωφέλεια. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιατί στα πλαίσια του ορισμού αυτών των υπηρεσιών η οδηγία αυτή δεν θα πρέπει να περιορίσει την ελευθερία των εθνικών υπηρεσιών, των περιφερειακών υπηρεσιών και των τοπικών υπηρεσιών να καθορίζουν οι ίδιες το τι είναι γενική ωφέλεια, κοινό συμφέρον κτλ. Σημαντικό επίσης και το άρθρο 2. Το άρθρο 2 αφορά τους ορισμούς. Εδώ ε, φαίνεται και η βασική αρχή του σημαντικού κινδύνου Τίθεται επίσης και το θέμα των κοινωνικών υπηρεσιών, δίδεται ιδιαίτερο βάρος στο θέμα των κοινωνικών υπηρεσιών, σημαντικότατο και το άρθρο 26 και αυτό γενικών αρχών είναι κάτι το οποίο έχει βρεθεί στο κέντρο πάρα πολλών διαπραγματεύσεων αναφέρεται εκτός από κοινωνικά κριτήρια και σε περιβαλλοντικά κριτήρια και λέγεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να σέβονται τις ε, εργατικές ρυθμίσεις οι οποίες ισχύουν σε κάθε χώρα, όπως επίσης και τις ε, νομικές ρυθμίσεις στον τομέα του περιβάλλοντος. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρχουν αντιθέσεις με αυτές. Τίθεται εδώ και το θέμα των ε, υπεργολαβιών μέσω διαγωνισμών <clears throat> και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Δόθηκαν αρκετές λεπτομέρειες από πλευράς του εισηγητή, δεν θα επανέλθω σε αυτές. Απλά θα πω ότι οι συμβιβαστικές του προτάσεις θα στηριχθούν σαφώς από μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω ορισμένες σκέψεις. Υπάρχουν ορισμένες πλευρές σημαντικές πάνω στις οποίες δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να ορίσουμε τον δρόμο που θα μας οδηγήσει καν στον συμβιβασμό. Καταρχάς, συνεργασία δημόσιου τομέα με ιδιωτικό τομέα και δεύτερον κάποιοι τομείς οι οποίοι λόγω του ειδικού τους χαρακτήρα χρήζουν εξαιρέσεων και αποκλήσεων. Έχουμε κάνει εδώ κάποια μικρά βήματα. Ελπίζω ότι η προσπάθεια η οποία θα συνεχιστεί στους τομείς αυτούς θα μπορέσει να μας επιτρέψει να καταλήξουμε θετικά και κυρίως να σεβαστούμε τη χρονική προθεσμία έτσι ώστε η συμβιβαστική αυτή πρόταση να ικανοποιήσει όλες τις πλευρές όσο αυτό είναι εφικτό. Επαναλαμβάνω η προσπάθεια του κυρίου Ζουβά είναι πολύ θετική. Τον ευχαριστώ για μια ακόμη φορά και ελπίζω τις επόμενες μέρες να μπορέσουμε να κλείσουμε το θέμα. Ευχαριστώ πολύ για την αισιοδοξία σας. Ο κύριος Χατζημαρκάκης τώρα, εξ του κύριου Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Εξ του κύριου Μπουσόη. Ο κύριος Μπουσόη ευχαριστεί την Επιτροπή για το σχέδιο οργανισμού και τον κύριο Ζουβέν για τις τροπολογίες που έχει προτείνει για να βελτιωθεί το κείμενο. Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από την οικονομική κρίση και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ε, δυνατότητα να επενδύουν οι μικροεπενδυτές στις χρηματαγορές. Θα πρέπει λοιπόν να αξιστεί η διαφάνεια και να υπάρχει ενημέρωση. Ο Κριστιαν Βουζό υποστηρίζει τις περισσότερες ε, ε, προτάσεις καθώς ε, στηρίζουν ε, την διαφάνεια όσον αφορά ε, τις δημόσιες συμβάσεις σε ζητήματα τεχνικών προδιαγραφών, ανάθεσης κτλ. Αλλά βεβαίως όπως έχει υποσχεθεί η Κομισιόν Προεκτή για ένα ελαφρύ ρυθμιστικό πλαίσιο. Επίση, χαίρεται ο κ. για το ότι βρήκαμε ένα καλό συμβασμό για την έννοια τη παραχώρηση, που βεβαίω έχει δημιουργήσει αρκετή νομολογία. Επίση, καλωσορίζει το νέο άρθρο για την αρχή τη ελεύθερη διοίκηση των δημοσίων αρχών, το οποίο σημαίνει πω μπορούν μόνε του να παρέχουν έργα ή υπηρεσίε ή μέσω μια παραχώρηση αναλόγω με το τι θεωρούν καλύτερο όσον αφορά τα κατόφλια. Και την μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αξίας της παραχώρησης είναι πάρα πολύ θετικό το ότι έχει εξορθολογιστεί το κείμενο και απλοποιηθεί. Ε, ο σχέδιος ηγητής της ε, Άλντε θεωρεί πως η αξία της παραχώρησης πρέπει να υπολογιστεί με βάση το συνολικό τζίρο ε, καθ' όλη τη διάρκεια της παραχώρησης ε, πλην φόρων. Συμφωνούμε βέβαια με το κατόφλι των ε, 2,5 εκατομμυρίων, αλλά δεν θεωρεί πως το κατόφλι πρέπει να φτάσει στα 8 ευρώ όπως προτείνει η Κομισιόν αντί για τα 5. Σε ε, αυτή την περίπτωση θα αποκλείσουμε πάρα πολλά συμβόλαια τα οποία σε άλλα κράτη-μέλη θα συμπεριλαμβάνονταν ε, εντός οδηγίας. Επιπλέον μπορεί αυτό να συγκρούεται με διεθνείς συμφωνίες τις οποίες έχει υπογράψει η Ένωση. Έχει επιτυχθεί επίσης ένας ικανοποιητικός συμβασμός όσον αφορά τον αποκλεισμό από το πεδίο εφαρμογή οδηγία. Έχουμε δηλαδή μια ισορροπημένη προσέγγιση και δεν έχει γίνει αυτή η οδηγία ένα που κάμισο αδιανό χωρί καμία περιορισμένη, χωρί καμία προσθέμενη αξία. Επίση σημαντικό είναι η εξαίρεση των ε, θηγατρικών και συνδεδεμένων επιχειρήσεων και οι εργασίες οι οποίες γίνονται εσωτερικά. Πρέπει όμως να ερμηνευθούν έτσι ώστε να μην υπάρχει άμεση, να μην υπάρχει στρέβλος του ανταγωνισμού μέσω της άμεσης ανάθεσης ε, σε δημόσιες ε, επιχειρήσεις οι οποίες θα βρίσκονται έτσι σε άμεσο ανταγωνισμό με την ιδιωτική αγορά. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε την απονομή τέτοιων ε, συμβάσεων παραχώρησης από αρχές οι οποίες δεν θα είναι οι αρχές ε, ε, οι οποίες ταυτόχρονα θα κάνουν την παραχώρηση και θα εκτελούν το έργο. Καθώς μην ξεχνάμε πως τα κριτήρια είναι πιο αυστηρά για εργασίες οι οποίες γίνονται από την ίδια την υπηρεσία. Επίσης θα πρέπει νομίζω να μείνουμε στο στο όριο του 19% για να μπορεί η ελεύθερη αρχή να λάβει αυτή την εξαίρεση. Επίσης, τα κριτήρια κοινού ελέγχου νομικού προσώπου, κ. Μπουζόη θεωρεί πω είναι σημαντικό να μην ε, επιδιώκουμε συμφέροντα τα οποία είναι διακριτά από αυτά της ελέγχουσας δημόσιας αρχής. Ακριβώς το συμφέρον είναι αυτό το οποίο ορίζει ε, το δημόσιο συμφέρον. να μιλάμε για αντικρώμενα συμφέροντα σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν δεν είναι σωστό. Ο κύριο Μπουσόη επίση καλωσορίζει τον συμβασμό για την διάρκεια τη παραχώρηση και ειδικά το ότι οι στόχοι απόδοση θα λαμβάνονται τώρα υπόψη ε, αν αν έχουμε επενδύσεις ή όχι. Η διατάξη για τη διαφάνεια και οι διαδικαστικές εγγυήσεις έχουν απλοποιηθεί κατά πολύ και υπάρχει τώρα μεγαλύτερος βαθμός ευελιξίας στις δημόσιες αρχές για την οργάνωση της διαδικασίας. Ε, πάντα με την εγγύηση της συμμεταχείρισης των υποψηφίων. Ο κ. είχε χαίρεται για το ότι είχε, έχει βρεθεί μια συμφωνία για την ε, ε, αξιολόγηση τεχνικών προδιαγραφών με βάση τεχνικές ή λειτουργικές απαιτήσεις. Και έτσι ενθαρρύνεται η καινοτομία. Τέλος, μια που μιλάμε για μακροχρόνιες συμβάσεις, όπου η αναδιαπραγμάτευση είναι μάλλον ο κανόνας, είναι σημαντικό να προβληθεί περισσότερη ευελιξία στην επαναδιαπραγμάτευση χωρίς μια νέα διαδικασία παραχώρησης. Επίσης ε, είναι σαφές ε, το τι είναι η ουσιαστική μεταβολή κατά οποία διευκολυνθεί η διαδικασία. Τέλος, θεωρούμε πως είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου τις σημαντικές βελτιώσεις που έχει επιφέρει ο εισηγητής μαζί με τους και εισηγητές. Ευχαριστώ. Um, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Χατζημαρκάκη, ε, προσωπήσα τον κύριο Μπουζόη. Λοιπόν, κύριε Αρούλε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Χάρμπορ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ζούμπα γιατί θα είναι αυτή η τελευταία μας συζήτηση, να τον ευχαριστήσω για την υπομονή του και για την ε, διάθεσή του πάντα να αναζητεί συμβασμούς και για την επαγγελματική του διεξαγωγή για την επαγγελματική διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων. Για να γίνει έτσι αυτή η πρόταση της Κομισιόν πιο απλή, να βρούμε καλύτερους ε, ορισμούς και ε, περισσότερη ευελιξία. Γι' αυτό νομίζω πως μπορούμε να δεχτούμε και να υποστηρίξουμε τους περισσότερους συμβασμούς. Όχι όλους, όμως πρέπει να διορθώσω τον κύριο Ζουβέν. Δεν θα δεχτούμε αυτές στο άρθρο 11 και 15 και τις μεταβατικές προθεσμίες. Παρ' όλα αυτά θέλω να τονίσω πως εμείς θα, προσπαθ... θα προτιμούσαμε να μην είχαμε τέτοια οδηγία. Αυτή η οδηγία θεωρούν πως θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσει. Αλλά οι θέσεις μας είναι γνωστές δεν θέλω να εξηγήσω το γιατί κάποιοι τομείς θα ήταν καλύτερο να αποκλειστούν. Μιλάμε για τις ε, υπηρεσίες γενικού ε, κοινωνικού συμφέροντος και τον τομέα των υδάτων. Δεν χρειάζεται νομίζω να πω περισσότερα. Τώρα θα το αποδεχτούμε αυτό. Έχει ευχαριστούμε τον κύριο Ζουβέν για το ότι ήταν διατεθειμένος να δει τι υπηρεσίε διάσωση ε, και καταστροφών. Αυτό το βρίσκουμε θετικό, αλλά τώρα να σας εξηγήσω το γιατί δεν θα μπορέσουμε να ε, υπερψηφίσουμε την έκθεση τελικά. Δυστυχώς θα πρέπει να την καταψηφίσουμε. Και το ζήτημα είναι εδώ πέρα η ε, συνεργασία. Γιατί εγώ διαφωνώ με τους προλαλήσαντες. Ε, δεδομένης της οικονομικής κρίσης θα πρέπει να εξυγχρονιστεί ο δημόσιος τομέας και να αναζητήσουμε συνέργειες. Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής υπάρχει κάτι το οποίο είναι σαφές πως μόνο μέσω συνεργασίας δημοσίων φορέων μπορούμε να επιτύχουμε συνέργεια έως και 30%. Αυτό χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή στα περισσότερα κράτη-μέλη και όχι μόνο λέμε γιατί μας λένε πως ε, το μέσο των υδάτων είναι μόνο γερμανικό ζήτημα. Όχι, σε πάρα πολλά κράτη-μέλη έχουμε δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες στην ίδια αγορά. Λίγα κράτη-μέλη είναι τελείως ιδιωτικά ή τελείως ε, δημόσια στον ε, τομέα αυτών. Τα περισσότερα έχουν μια μεικτή εικόνα. Θα πρέπει λοιπόν να μπορεί να εργαστεί λογικά ο δημόσιος τομέας. Βεβαίως χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες, βεβαίως πρέπει να τηρήσουμε τις αποφάσεις του ΔΕΚ, για ζητήματα ιδιωτικής συμμετοχής, ε, για τα ζητήματα τα οποία είναι ουσιαστικά για την παροχή των υπηρεσιών, για το ποιος θα ασκεί τον έλεγχο, αλλά το ζήτημα είναι ο ορισμός και θεωρώ πως ο ορισμός του κριτηρίου της ουσιαστικής υπηρεσίας υπήρχε ήδη στην έκθεση Ταραμπέλα και εδώ πέρα έγινε ακόμη ε, καλύτερος. Οπότε, λόγω αυτής της ε, αλλαγής ε, εδώ πέρα, ενώ απήχαμε στην έκθεση Τραμπέλα θα πρέπει να καταψηφίσουμε. Μην ξεχνάμε πως 80... Όταν ε, ένα 80% των ε, εσόδων πηγαίνει σε ένα δημόσιο φόρεα, υπάρχει ένα πρόβλημα γιατί το ζήτημα αφορά και τον τομέα των υδάτων και τη ενέργεια. Αλλά βεβαίως ο τομέας τη ενέργειας έχει απελευθερωθεί, υπάρχουν υποχρεώσει για να γίνει κάποιος διαγωνισμός, αλλά τι θα γίνει. Θα οδηγηθούμε τότε, όταν συμψηφίζουμε τους τομείς ενέργειας και υδάτων και σε πλήρη ιδιωτικοποίηση του τομέα υδάτων. Και αυτό είναι δυσκολία γιατί και το νερό πρέπει να έχει συγχρονιστεί, δηλαδή η παροχή υδάτων, η αποχέτευση και εκεί πέρα να υπάρξουν συνέργειες και πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν και οι περιφερειακοί δήμοι ε, μεγάλη και μικρή και χρειάζεται μια καλύτερη μέθοδος για να τους καλύψουμε και αυτούς. Ε, με αυτό είναι εδώ πέρα την πρόταση όλα αυτά κινδυνεύουν. Η οδηγία αυτή δεν απαιτεί βεβαίως την ιδιωτικοποίηση του τομέα της ίδρυψης. Αλλά τι θα γίνει. Θα δυσκολευτούν οι Δήμοι να τηρήσουν τους όρους και άρα θα βρεθούμε σε μια αβεβαιότητα νομική και μετά θα σκεφτούν οι Δήμοι μήπως καλύτερα να το ξεφορτωθούμε το νερό για να αποφύγουμε δικαστικές περιπέτειες. Και αυτό είναι το πρόβλημα, γι' αυτό θα καταψηφίσουμε αυτή την οδηγία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Good, thank you very much. Just... Uh, Ευχαριστώ πολύ. Κάποια σύντομα πράγματα σαν σκιώδης εισηγητής, όχι σαν πρόεδρος. Έχω ασχοληθεί με το θέμα μέσω των υπολείπων οδηγιών για τις δημόσιες προμήθειες. Εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα στη γραμμή του κυρίου Ζουβά. Χρειάστηκε βέβαια να κάνουμε κάποιες βασικές αλλαγές στην αρχική πρόταση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε σε επίπεδο προστιθέμενης αξίας στην αρχική πρόταση. Κάτι τέτοιο είχε προκαλέσει αρκετές αμφιβολίες. Ελπίζω αυτό να βοηθήσει. Θα μπορέσουμε έτσι να ενθαρρύνουμε τις εξελίξεις στον τομέα αυτό των παραχωρήσεων, των συμβάσεων παραχώρησης. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Η φύση βέβαια των παραχωρήσεων είναι τέτοια που απαιτεί περίπλοκες ρυθμίσεις απαιτεί περίπλοκες συμφωνίες, έχουν μακρά διάρκεια, υπόκεινται σε μακρόχρονες διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία αυτού που αναλαμβάνει την παραχώρηση και η προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις σε επίπεδο τεχνολογίας και σε άλλους τομείς περιβαλλοντικούς κτλ. Υπάρχει επίσης και πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία τύπων παραχωρήσεων τέτοιων συμβάσεων παραχωρήσεις. Και δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε μη ρεαλιστικούς περιορισμούς. Κατανοώ την ευαισθησία για κάποιους τομείς, αναφέρθηκε σε αυτούς η κυρία Ρούλε, αλλά υπάρχουν χώρες τις οποίες υπάρχουν συμβάσεις παραχώρησης και για την εκμετάλλευση ε, και διάθεση του ύδατος. Είμαστε ικανοποιημένοι λοιπόν από την προσπάθεια του κυρίου Ζουβά. Έχουμε ένα καλό πακέτο πλέον μπροστά μας. Θα πρέπει να δούμε τι θα μείνει από αυτό μετά την ψηφοφορία. Να δούμε αν κάποια στοιχεία δεν είναι απαραίτητα, δεν είναι τα καλύτερα, δεν συνεισφέρουν στην απλοποίηση. Αλλά αυτό φυσικά αφορά λεπτομέρειες και όχι την ουσία της πρότασης και θα πρέπει να σεβαστούμε και τα όρια τα οποία προτείνει η συγκεκριμένη αυτή προσπάθεια. Η κυρία Σιχόφσκα είναι εδώ. Α, όχι. Έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει η κυρία Φερχαέν. Να ευχαριστήσω και εγώ τους συναδέλφους ε, και τον κύριο Ζουβέν για την καλή συνεργασία. Τα άρθρα 11 και 15 εμείς ε, ως ε, απλά μέλη της Επιτροπής ε, τα ελάβαμε μόλις χτες, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε τις λεπτομερείς διαπραγματεύσεις. Οπότε θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτον, κάτι γι' αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κατσιμαρκάκης εξ ονόματος του κ. Μπουζό. Είναι σημαντικό, αν και Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το επίπεδο των μισθών, παραδείγματο χάρη, και άρα το κατόφλι μετά που προκύπτει, ε, αυτό το πρόβλημα ισχύει γενικώ. Εκεί, ε, γιατί οι υπηρεσίες βεβαίως είναι υπηρεσίες έντασης εργασίας ε, και κάποιες συμβάσεις σε μια χώρα θα είναι κάτω από το κατόφλι, ενώ σε άλλες ε, πάνω από το κατόφλι. Οπότε δεν νομίζω πως είναι πολύ βάσιμο αυτό το επιχείρημα. Νομίζω πως μπορούμε να ορίσουμε ένα ενιαίο κατόφλι. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο είπε η Χάιντερ για την συνεργασία των Δήμων. Νομίζω ειδικά ε, λόγω της κρίσης και του στόχου που ακολουθούμε όλοι, ε, πρέπει να χρησιμοποιούμε το χρήμα των φορολογουμένων ε, αποτελεσματικά. Και ο δημόσιος τομέας πρέπει να έχει κάθε δυνατότητα να το κάνει. Και να μην του βάζουμε μόνο προσκόμματα. Για να μην μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Οπότε αναμένω το κείμενο για το άρθρο για τη συνεργασία των Δήμων. Τώρα, για τις ε, θηγατρικές υφιστάμενες επιχειρήσεις ε, ή την ε, εσωτερική εκτέλεση κάποιων έργων. Δεν ξέρω τι εννοεί εδώ πέρα το κείμενο, αλλά σίγουρα θα υπάρξουν διαφορετικές ερμηνείες στα κράτη-μέλη. Εμείς μην ξεχνάμε πως υπάρχουν ε, δημοτικές ε, επιχειρήσεις ε, οι οποίες όμως ελέγχουν και το νερό και το ρεύμα και δεν αποκλείονται άρα 100% από την οδηγία όπως λέμε πάντα γιατί υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες όσον αφορά τον κανόνα αυτού, αυτό του 80-20 στον απελευθερωμένο δηλαδή τομέα της ενέργειας ε, όπου παρέχονται υπηρεσίες. Οπότε θα ήθελα εγώ μία διευκρίνηση σε μία συμβαστική λύση, δηλαδή όπου οι δημοτικές επιχειρήσεις ε, δραστηριοποιούνται και οι υπηρεσίες τους παρέχονται 100% εντός του Δήμου και είναι τοπική επιχείρηση, ε, να εξαιρεθούν από την οδηγία. Uh, uh, Ευχαριστούμε κύριε Βερχέιν. Ξέρω πόσο αφοσιωμένοι είστε στο θέμα αυτό. Σας ε, ευχαριστώ θερμά για τη συμβολή στη συζήτηση. Ε, δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο. Κυρία Σικόφσκα, παρακαλώ εν συντομία γιατί περιμένουν οι καλεσμένοι μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ σας εύχομαι καλή χρονιά και από το την ομάδα για τις συμβάσεις παραχώρησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και και τον εισηγητή για το μέχρι τώρα έργο και εκτιμούμε ιδιαίτερα την πρόοδο που έχει συντελεστεί. Όπως είπα και στο παρελθόν, θεωρούμε ότι όντως το κείμενο απλοποιήθηκε αισθητά. Πάντως οι βασικές αρχές και η λογική της πρότασης έχουν διαφυλαχθεί και χαιρόμαστε ιδιαίτερως γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά έχω τέσσερα σχόλια σημαντικά κατά τη γνώμη μου. Γιατί δεν θα είναι άμερα συνεπειών. Καταρχήν, πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Προσθέθηκαν ε, και άλλες εξαιρεσει από την οδηγία εφαρμογή. Καταρχήν, τα ε, τυχερά παιχνίδια. Θεωρούμε ότι δύσκολο μπορούμε να τεκμηριώσουμε ε, να δικαιολογήσουμε μια τέτοια εξαίρεση. Βέβαια προσπάθησαν ε, να επιχειρηματολογήσουν σχετικά. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της εξαίρεσης των τυχερών παιχνιδιών του τζόγου. Επίσης δεν θεωρούμε ότι έχει νόημα να εξαιρεθούν ε, το δραστηριότητες στο, στα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχουν ούτε νομικές ούτε οικονομικές αιτίε και λόγοι για να δικαιολογούνται τέτοιε εξαιρέσει. Βέβαια, για κάθε δραστηριότητα ισχύουν στου διαφορετικέ νομοθετικέ διατάξει, αλλά ακριβώ ο στόχο τη οδηγία είναι να προσφέρει έναν ελάχιστο κοινό παρανομαστή. Γιατί τέτοιου είδου ε, ε, ετερόκλητε πρακτικέ δεν συνάδουν με τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση πάντα. Τρίτο θέμα, τα κατόφλια. Όπω ακούσαμε και στη συζήτηση, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι διεθνεί μα υποχρεώσει και ιδιαίτερα το GPA. Οποιαδήποτε απόκληση από τις υποχρεώσεις αυτές θα έχει σημαντική επίδραση στη σχέση μας με τις τρίτες χώρες. Για το άρθρο 15 θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη των επιχειρήσεων μεταξύ κρατικών αρχών, αλλά όπως φάνηκε και από την ομολογία του ΔΕΚ, σε ιδιαίτερα, ε, σε, ιδιαίτερα θέματα συμμετοχής του ιδιωτικού κλάδου ε, δεν είναι δυνατή η ε, σύναψη μόνο μεταξύ δημοσίων. Θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη. Τώρα, για τα κριτήρια και τις διαδικασίες της ανάθεσης. Ε, ίσως είναι θέμα διατύπωσης, αλλά μια και το σχετικό άρθρο έχει αναδιατυπωθεί, με σημαντική αλλαγή του περιεχομένου, φοβόμαστε μήπως υπάρξει διακριτική μεταχείριση μεταξύ κάποιων υποψηφίων λόγω διαδικασίας. Ελπίζω στη συζήτηση να διευκρινιστούν αυτά τα σημεία στη συνέχεια. Πάντως, επαναλαμβάνω ότι εκτιμούμε ιδιαίτερο στην πρόοδο που έχει γίνει μέχρι στιγμής και είμαστε στη διάθεση της Επιτροπής σα για περαιτέρω συζητήσεις. Ευχαριστούμε. Πράγματι, τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας είναι ορατά πλέον. Κύριε Ζουβά, θα θέλατε να κλείσετε τη συζήτηση. Σύντομα κύριε Πρόεδρε, όλοι εκφράστηκαν, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές εκτιμήσεων ανάμεσα στους βουλευτές, ανάμεσα σε εμά και στην Επίτροπη, αυτό είναι το παιχνίδι της δημοκρατίας εφόσον το Κοινοβούλιο δεχθεί το κείμενο και το εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για αυτό που κάνουμε. Εμείς κάνουμε βιώσιμη, καθιστούμε βιώσιμη την κοινοβουλευτική δημοκρατία μέσω της δημιουργίας ενός νομοθετικού κειμένου. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κ. Μπάρμπορ. Να σας θυμίσω ότι η ψηφοφορία θα, είναι, θα γίνει την 24η Ιανουαρίου. Θα υπάρξουν πάρα πολύ εντατικές ψηφοφορίες εκείνη την ημέρα. Και για όλα αυτά τα θέματα η τελευταία λέξη θα υποθεί την επόμενη εβδομάδα. Περνάμε τώρα στις συζητήσεις με συνεισφορές από διάφορους εμπειρογνώμονες σε δύο γνωμοδοτήσεις τις οποίες ε, εκφέρουμε προς την Οικονομική Επιτροπή σχετικά με τις καταναλωτικές πλευρές δύο πολύ σημαντικών προτάσεων. Καταρχάς, βασικές κομβικές πληροφορίες για επενδυτικά προϊόντα. Συντάκτης μας είναι ο κύριος Παντσέρη, τον οποίο ήδη ακούσαμε σήμερα, ο σκληρά εργαζόμενος. Και δεύτερον είναι η νέα πρόταση για ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Έχουμε κάνει προσπάθειες στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα στο θέμα των επενδυτικών προϊόντων, όπως επίσης και στο θέμα των στεγαστικών προϊόντων και συνεπώς καταφέραμε να συγκεντρώσουμε τέσσερις εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα μας μεταφέρουν τις δικές τους προοπτικές για τα θέματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε στα πλαίσια της πρότασης που θα κάνουμε προς την Οικονομική Επιτροπή. Είμαστε σε συζητήσεις με την Οικονομική Επιτροπή για το αν θα υπάρξει μια σύνδεση των Επιτροπών Οπότε κάποιες από τις τροπολογίες ε, θα υποχρεωθούν να τις δεχθούν δικές μας, αλλά αυτό είναι ένα θέμα πολιτικό αστηρά και οι συζητήσεις ε, ε, για μια συμφωνία με την Οικονομική Επιτροπή συνεχίζονται. Έχουμε δύο λοιπόν προτάσεις μπροστά μας. Θα ήθελα να μου πούνε οι συγητές το πώς πιστεύουν ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε. Πρότασή μου θα ήταν πρώτα να ακούσουμε μια εισαγωγή από τον κύριο Παντζέρη για ε, τις βασικές λεγόμενες πληροφορίες και μετά να ακούσουμε τους δύο εμπειρογνώμονες για τον κλάδο αυτό, τον κύριο Σαβιανό και τον κύριο Πουρκάτη αν ακούσαμε καλά, μετά από την παρέμβαση του κυρίου Παντζέρη και θα υπάρξουν αμέσως μετά κάποιες ερωτήσεις και σχόλια από τους Σκιώδης. Έχουμε λίγο καθυστερήσει, θα προσπαθήσουμε να μοιράσουμε το χρόνο που έχουμε στις δύο αυτές εκθέσεις. Και μετά θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Στήλερ, η οποία είναι η συγγήτριά μας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και θα ακούσουμε τον κύριο Όξλι και την κυρία Κόλερα που είναι οι δύο εμπειρογνώμονες. Θα σας καθοδηγούμε σχετικά με τις χρονικές προθεσμίες. Μετά θα ακούσουμε τα μέλη και θα ακολουθήσει διάλογος ανάλογα με το χρόνο. Κάτι διαδικαστικό. Μια ερώτηση λέει ο κύριος Μπιερνό. Θα έχουμε τη δυνατότητα να εκφράσουμε και την γνώμη μας για τους καταναλωτές. Θα ήθελα, εν πάση περιπτώσει, και για την πρώτη οδηγία να προσπαθήσω να εκφράσω κάποιες απόψεις, λέει ένας από τους εμπειρογνώμονες. Δεν ξέρω αν θέλετε να αντιστρέψουμε τη σειρά. ο κύριος Κάρτη. Και εγώ θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για το IMD. Ε, δεν ξέρω, εξαρτάται από σας. Κοιτάξτε, έχουμε κάποιο χρόνο για να επωφεληθούμε από την παρουσία σας εδώ. Αν ακολουθήσουμε λοιπόν την πρότασή μου, νομίζω ότι και οι τέσσερις μπορείτε να σχολιάσετε όλες τις παρεμβάσεις σας. Είμαστε ευέλικτοι και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε σωστά την παρουσία σας ανάμεσά μας. Και από, το όπως γνωρίζετε μπορείτε να ομιλήσετε ή αδίποτε γλώσσα επιθυμείτε. Υπάρχει πλήρης διερμηνευτική υπηρεσία. Και οι σκιώδεις θα μιλήσουν μετά τους εμπειρογνώμονες. Δεν ξέρω ποιοι σκιώδεις είναι εδώ, η κυρία Ρούλε είναι εδώ και για τις δύο οδηγίες ο κύριος Καράς, τον οποίο καλωσορίζω, ο οποίος είναι απασχολημένος συνομιλώντας με μία συνάδελφο. Είναι σημαντικό μέλος και της Οικονομικής Επιτροπής. Με χαρά σας βρίσκουμε στην Επιτροπή μας. Δεν βλέπω ελευθέρους. Η κυρία Χάντσλεκ επίσης είναι παρούσα, η οποία αντικαθιστά την κυρία Πιετικάινεν. Υπάρχουν άλλες αντικαταστάσεις. Ε, λοιπόν, ε, πέρα από τα εισαγωγικά, τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Παντσέρη για να κάνει μια σύντομη εισαγωγή στην πρότασή του. Και μετά θα περάσουμε το λόγο στους εμπειρογνώμονες, με τον κύριο Μπιερνό πρώτο. Ο κύριος Παντσέρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πριν μπω στην ουσία της έκθεσης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι χθε κατατέθηκε η αναθεωρημένη πρόταση. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη από εδώ και πέρα. Ε, προς το παρόν έχουμε την πρόταση αυτή μόνο στα αγγλικά γιατί δεν μπορέσαμε λόγω των διακοπών να έχουμε τις άλλες μεταφράσεις οι οποίες θα είναι μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου διαθέσιμες. Το δεύτερο θέμα το οποίο ήδη θέσατε εσείς και το οποίο πολιτικά θα έλεγα απαιτεί την ενισχυμένη συνεργασία με την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Θα πρέπει να διευκρινιστεί το θέμα αυτό έτσι ώστε να μπορέσουμε να εργαστούμε με σοβαρότητα και ηρεμία. Επί της ουσίας θα πρέπει να δεχτούμε θα έλεγα ευνοϊκά την πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την σχετική με τις βασικές ενημερωτικές και ε, ε, πληροφορίες μάλλον που περιλαμβάνονται ε, στους φακέλους των επενδυτικών προϊόντων. Ο καταναλωτής που θέλει να χρησιμοποιήσει τέτοιες υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει το τι σημαίνουν και να μπορεί να συγκρίνει. Αυτές ε, οι προσυμβατικές αν θέλετε πληροφορίες πολλές φορές είναι εκπεφασμένες με ιδιαίτερα τεχνικό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τίνει στη δημιουργία ενός ε, προτύπου θα έλεγα καθορισμένου το οποίο θα καλύψει κάποια έλλειψη που παρατηρείται στη σωστή ενημέρωση του καταναλωτή επενδυτικών προϊόντων να μπορέσει να βρει τα επενδυτικά προϊόντα γνωρίζοντας το περιεχόμενό τους. Υπάρχουν αρκετές λοιπόν θετικές προτάσεις ε, στην πρόταση. Στόχος είναι να καταστούν οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες, κατανοητές, με απλή γλώσσα σε κομβικά κεντρικά θέματα. Δεύτερον, να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων μέσα από ένα εναρμονισμένο πλαίσιο παρουσίασης των επενδυτικών προτάσεων. Τρίτον, υποχρέωση παροχής κομβικών πληροφοριών στον καταναλωτή πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Και τέλος, επιβολή κυρώσεων, ένα καθιστός επιβολής κυρώσεων στην περίπτωση κατά την οποία ο κανονισμός δεν γίνεται σεβαστός. Νομίζω ότι μία σειρά προτάσεων θα πρέπει να βελτιωθεί και να συμπεριληφθεί στην προτινόμενη έκθεση χωρίς να μπω επί της ουσίας θα αναφερθώ σε κάποιες από αυτές τις ρυθμίσεις. Καταρχάς δεν θα πρέπει να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου κανονισμού. Οι εξηγήσει θα πρέπει να δίδονται όχι μόνο από τους παροχείς των συγκεκριμένων προϊόντων αλλά και από τους ενδιαμέσους. Δεν θα πρέπει να περιορίζονται σε αυστήρα επενδυτικά προϊόντα αλλά και σε μεικτά προϊόντα τα οποία είναι γνωστής απόδοσης θα πρέπει επίσης να καλύψουμε και κάποια συνταξιοδοτικά επιχειρηματικά συστήματα. Οι εξηγήσει και παρουσιάσεις των κινδύνων δεν θα πρέπει να περιορίζονται ε, στις ε, ρυθμίσεις που ισχύουν για τις επενδύσεις στον τομέα των στεγαστικών και θα πρέπει οι εξηγήσει αυτές να δίδονται στον καταναλωτή τη στιγμή κατά την οποία γίνεται η πρόταση από τον ε, επιχειρηματία το πιστοτικό ίδρυμα ή κάτι άλλο. Και θα πρέπει να έχουν ε, λοιπόν παρουσιαστεί στον καταναλωτή όλες αυτές οι εξηγήσει ακόμα και για προϊόντα με τα οποία δεν θα, ε, για τα οποία δεν θα προηγηθεί άμεση επαφή. Είναι απαραίτητο όμως να ε, υπάρξει πλήρης ενημέρωση ακόμα και με ηλεκτρονικό τρόπο. Για λόγους συντακτικούς δεν μπορέσαμε να καλύψουμε πλήρως όλους τους τομείς, θα πρέπει να υπάρξει μια τροπολόγηση της πρότασης σχετικά με τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την παροχή πληροφοριών και σχετικά με τη σωστή ενημέρωση των καταναλωτών σε επίπεδο διαφημίσεων. Εδώ έχουν ε, γίνει ορισμένες ρυθμίσεις και για τις λεγόμενες εναλλακτικές δυνατότητες επίλυσης διαφορών. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει δεκτό. Ε, θα έλεγα ότι έχουμε ένα σημαντικό πακέτο μπροστά μας και θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με τους σκιώδεις εισηγητές έτσι ώστε να καταλήξουμε σε επιθυμητές λύσεις. Έχουμε λοιπόν μια πρώτη δυνατότητα ε, σύγκρισης των ε, ιδεών ε, και έβρεσης των απαιτούμενων λύσεων. Ευχαριστώ. Πράγματι είχαμε και το σχέδιο γνωμοδότησή σα που αποτέλεσε μια πάρα πολύ καλή βάση για τις συζητήσεις και για τις συζητήσεις με την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών. Η αρχική απάντηση του Προέδρου της Επιτροπής αυτής στο αίτημα μας ήταν μια ξεκάθαρη άρνηση ε, και μας είπε πως οι συζητήσεις συνεχίζονται, αλλά νομίζω τελικά πως η διάσκεψη των Προέδρων, ε, ο Πρόεδρος, ο κύριος ε, θα πρέπει να λάβει μια απόφαση. Προχωράμε. Λοιπόν, χαίρομαι που καλωσορίζω τον Ζαν Φρανσουά τον πρώτο μας εμπειρογνώμονα. Έχετε νομίζω τα βιογραφικά τους, των ειδικών. Θα ήθελα λοιπόν να τον καλωσορίσω ιδιαίτερα γιατί θα μας παρουσιάσει εξ ονόματος του Μπιούκ που βεβαίω είναι συχνά στις συναντήσεις μας και επειδή έχει και εμπειρία συμβουλών στο τεστ ΑΣΑ, ένα βελγικό Ινστιτούτο Συγκρίσεων Καταναλωτικών Προϊόντων. Ε, σας δίνω λοιπόν τον λόγο για 10 λεπτά το πολύ για την πρώτη σας ε, παρέμβαση, ειδικά ε, όσον αφορά αυτά τα έγγραφα πληροφόρησης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την εισαγωγή σας αυτή. Θα συνεχίσω στα γαλλικά. Για τα αρχικά και για δεν είναι, όσοι δεν είναι εξοικειωμένη. Το KID είναι τα βασικά, βασικές πληροφορίες σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα. Επίσης τα PRIX Package είναι κάποια επενδυτικά προϊόντα. Και σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να δούμε αν θα πρέπει να ισχύει μόνο για, τις τα συγκεκριμένα πακέτα επενδύσεων ή να, επεκτείνεται και σε άλλες επενδύσεις ε, αποταμίευσης. Σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι μια πρωτοβουλία που την περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό και τη χαιρετίζουμε έθερμα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα σύντομο έγγραφο με συγκεκριμένα σαφή και ευανάγνωστα για τους καταναλωτές σημεία. Και μάλιστα αυτό φάνηκε και σε ε, μελέτες για την συμπεριφερολογική οικονομία. Σημαντική ε, μελέτη που έδειξε ότι τα ΒΕΠ, οι βασικές πληροφορίες για τα περιοδικά προϊόντα είναι θεμελιώδη σημασία για του καταναλωτέ για να μπορούν να, ε, να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή. Για μας όλα τα προϊόντα αποταμιεύση και επένδυση θα πρέπει να έχουν μια, ένα, ένα είδους για τις βασικές πληροφορίες και να καλύπτονται οι, οι βασικές ερωτήσεις και προβληματισμοί. Το άρθρο 8. Χρειάζονται απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές για όλα τα προϊόντα πριν κάποιος λάβει μια απόφαση. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την ιδέα, το KID, οι βασικές πληροφορίες, το web, να γενικευθεί. Σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα με τις βασικές πληροφορίες, αυτό που λείπει από την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάποιες πληροφορίες που δίνει μόνο ο διανομέας. <clears throat> Σε ό,τι αφορά το κόστος, τα έξοδα, όταν, κανείς, όταν κάποιος επενδύει σε ένα προϊόν. Τα έγγραφα με τις βασικές πληροφορίες του εκδότη αναφέρουν τα πιο υψηλά έξοδα, το μεγαλύτερο κόστος που μπορεί να απαιτηθεί στο πιο δαπανηρό διάβολο διανομής. Αν ο καταναλωτή στηριχθεί στα πιο ακριβά τέλη που προβλέπει το έγγραφο με βασικές πληροφορίες τη Επιτροπής θα παραμερίσει κάποιε άλλες επενδύσεις που μπορεί να είναι πιο ενδιαφέρουσε. γιατί ο μεσολαβητή του εξασφαλίζει μια επιστροφή ο μεσάζων ή αν στραφεί σε διαφορετικό διάβλο διανομή, έχει πολύ χαμηλότερα ε, έξοδα από αυτά που αναφέρονται. Οπότε αυτό που ζητούμε είναι ο μεσάζων σε ένα παράρτημα ίσως ε, στο έγγραφο με τις βασικές πληροφορίες να αναφέρεται το πραγματικό κόστος που θα πληρώσει κανείς όταν περνάει από μεσάζοντα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι η φορολογία του προϊόντος. Τα πρίψ που λέμε, αυτές οι έμεσες επενδύσεις που είναι packaged, είναι κάπως προκαθορισμένες και περιλαμβάνονται στο πακέτο είναι διαφορετικά. Μπορεί να έχουμε μια διαρθρωμένη επένδυση, ένα ασφαλιστικό προϊόν, ένα οσεκά και ούτω καθεξής. Για όλα αυτά τα προϊόντα έχει διαφορετικές φορολογικές διατάξεις. Οπότε αν κανείς κάνει την επιλογή του χωρίς να λάβει υπόψη και τη φορολογία, θα κάνει λάθος την επιλογή, δεν θα επιλέξει το καταλληλότερο προϊόν. Γι' αυτό και μια σύντομη ενημέρωση και για το φορολογικό καθεστώς είναι απαραίτητη. Και μόνο ο διανομέας μπορεί να τη δώσει, γιατί ο εκδότης δεν ξέρει σε ποια χώρα θα κυκλοφορήσουν αυτά τα προϊόντα. Οπότε, καλό θα ήταν ο διανομέας να συμπεριλαμβάνει ένα παράρτημα με το ακριβές κόστος, το πραγματικό κόστος, το φορολογικό καθεστώς και επίσης ε, οι υποχρεωτικές πληροφορίες που θεσπίζονται στη Μηφίτη, για παράδειγμα στην οδηγία ε, να συμπεριλαμβάνονται σε ένα ενιαίο έγγραφο και να μην είναι κατακαιρματισμένες. Βέβαια θα είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί αυτός ο κανονισμός ως κατεξουσιδότηση πράξη για τη ΜΥΦΙΤ. Αλλά αν τα δούμε όλα υπό το πρίσμα του καταναλωτή, νομίζω ότι είναι σκόπιμο όλες οι πληροφορίες αυτές να περιλαμβάνονται σε ένα και μόνο έγγραφο, για να γίνει δυνατή η σύγκριση μεταξύ των διαφόρων επενδυτικών προϊόντων. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση και τις πληροφορίες για τον κίνδυνο στο έγγραφο με τις βασικές πληροφορίες για, τα, για τις ΟΣΕΚΑ έχουμε μία κλίμακα από 1 έως 7 ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου. Δεν είναι το καλύτερο σύστημα, αλλά για, τα για το σωσικά αρκεί. Αλλά και για τα άλλα πακέτα τα επενδυτικά ισχύουν διαφορετικοί κίνδυνοι γιατί στους ΟΣΕΚΑ έχουμε αναγκαστικά μια διαφοροποίηση, δηλαδή διαφορετικά προϊόντα στον ίδιο ΟΣΕΚΑ. Ενώ ε, μπορεί να έχουμε ένα ασφαλιστικό προϊόν με unit link και επένδυση σε ένα προϊόν. Εκεί ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος σε περίπτωση πτώχευσης του εκδότη, του συγκεκριμένου προϊόντος. Οπότε δεδομένη τη διαφοροποίηση των κινδύνων, θα πρέπει να δούμε πώ θα ενημερώσουμε καλύτερα τον καταναλωτή. Κάτι που παραλείπεται αυτή τη στιγμή από την πρόταση τη Επιτροπή. Αυτό που ζητούμε είναι οι ευρωπαϊκέ εποπτικέ αρχέ, ΕΣΜΑ, ΙΟΠΑ, EBA, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, να εγγύψουν στο θέμα αυτό και να αναλύσουν τις διάφορες δυνατότητες ενημέρωσης και να δουν ποια είναι η καταλληλότερη ενημέρωση για τους καταναλωτές. Αυτή η μεθοδολογία χρησιμοποιώθηκε για τα έγγραφα με βασικές πληροφορίες για το ΣΟΣΕΚΑ και την ίδια μέθοδο που θεωρούμε εξαιρετική ε, ζητούμε να την εφαρμόσει η Επιτροπή και στην περίπτωση αυτή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξαίρεση, το έγγραφο με τις βασικές πληροφορίες θα πρέπει να δοθεί από τον ε, μεσάζοντα πριν την συνδιαλλαγή προβλέπει ο κανονισμός. Όχι δηλαδή ότι όταν δίνεται απλώς μια συμβουλή χωρίς διαλλαγή. Θα πρέπει να δοθούν αυτά τα έγγραφα με βασικές πληροφορίες πριν τη συνδιαλλαγή. Προβλέπεται όμως η δυνατότητα να μην δοθούν τέτοιε πληροφορίες όταν έχουμε εξ αποστάσεως ε, επαφή και όταν δίνεται η, εντολή, η επενδυτική εντολή. Υπάρχει ένα κενό πολύ σημαντικό που καλό θα ήταν να έρθει γιατί αλλιώ οι διανομή, οι τράπεζε. που επιτελούν αυτή τη ε, λειτουργία, θα προτιμήσουν τις τηλεφωνικές συνομιλίες για την παροχή συμβουλών, αντί να στέλνουν τα έγγραφα, κάτι που απαιτείται για την ε, πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση. Αυτά ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστώ θερμά. Πολύ εμπεριστατωμένη η ενημέρωση και βλέπω ότι συμφωνείτε σε πολλά σημεία και με τον εισηγητή μας, τον κύριο Παντζέρη. Περνάμε τώρα στον επόμενο μας καλεσμένο για το ίδιο θέμα, τον κύριο Πολ Κάρτη, που έχει πλούσια πείρα στις ασφαλίσεις, στις ασφάλειες μάλλον, και θα ήθελα να δώσω το λόγο για να σχολιάσω το δεύτερο θέμα, την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Ο κύριος Κάρτη είναι πρόεδρος Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας ε, ε πολιτικών διαμεσολαβητών και του δίνω το λόγο για ένα δεκάλεπτο. Το πολύ. Thank you very much, um, chairman. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα φροντίσω τα σύντομα μου να είναι σχόλια γιατί με την άδειά σα θα ήθελα εγώ να παρέμβω στο κομμάτι IMD. Οπότε, ε, δέκα λεπτά επί τέσσερις ανθρώπους επί θα φτάνουμε στα 80. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Στάιλερ και τον κύριο Παντσέρη που μας προσκάλεσαν εδώ να κάνουν μια παρουσίαση και θα κάνω και εγώ κάποιες ε, παρεμβάσεις. Να πω πρώτα απ' όλα ποιος είμαι, για όσους ίσως ε, δεν το ξέρουν. Και μετά θα προσπαθήσω να κάνω μια σύνοψη. Πρώτα απ' όλα, για όσους δεν το ξέρουμε εμείς, εκπροσωπούμε τους ενδιάμεσους ε, στην Ευρώπη. Έχουμε 50 ενώσεις μέλη και εκπροσωπούμε άνω του ενός εκατομμυρίου ε, ενδιαμέσων, η συντριπτική των οποίων είναι σχετικά μικρές επιχειρήσεις και βρίσκονται σε κάθε γωνία της Ένωσης και είναι η πιο άμεση επαφή των καταναλωτών. Οπότε μαζί με τους καταναλωτές ε, εμείς είμαστε αυτοί που αγγίζει περισσότερο αυτή η πρόταση. Επίσης, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το ότι έχουμε μια πολύ, πολύ ανταγωνιστική αγορά, που δεν υπάρχει μόνο ενδιάμεση, αλλά πάρα πολλές άλλες μορφές και διάβλη διανομής, που συνεχώς ανταγωνίζονται για τους ε, πελάτες τους και πρέπει να αντιληφθούμε πως είναι πολύ ανταγωνιστική η αγορά και να αντιληφθούμε πως όποιες προτάσεις γίνουν ε, μπορούν να διαταράξουν αυτή τη δυναμική ίσως και για το χειρότερο. Αυτό ως ένα γενικό σχόλιο. Το δεύτερο γενικό σχόλιο θα ήθελα να κάνω το εξής βεβαίως οι ασφαλείς έχουν τις ιδιαιτερότητές τους που δεν μπορούμε να ξεχνάμε. Οπωσδήποτε υπάρχει εδώ πέρα περιθώριο για τυποποίηση προς το συμφέρον των καναλτών. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτό, αλλά υπάρχουν ιδιαιτερότητες που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Σε σχέση με τα πρίψη. Συμφωνώ πλήρως με τα σχόλια του κυρίου Παντσέρη πως πρέπει το έγγραφο πληροφοριών να είναι αξιόπιστο, συγκρίσιμο και προφανώ να έχει και κάποιο νόημα. Το μέτρο δυνατού πρέπει να είναι και τυποποιημένο και συμφωνούμε βεβαίως πώς θα πρέπει να να υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες. Επίσης, προφανώς κάποια εναρμόνιση και όλες αυτές τις πληροφορίες ε, να δίνονται πριν από την σύναψη της σύμβασης. Αυτό εξυπακούεται. Έχουμε κάποια προβλήματα όμως με τις απόψεις ε, που ακούγονται. Ένα είναι πως θεωρούμε πως το να είναι συνυπεύθυνοι η ενδιάμεση με τον παραγωγό είναι επικίνδυνο. Δημιουργεί έτσι, εάν είναι δύο ε, μέρη συνυπεύθυνα, η δυνατότητα νομικής αβεβαιότητας που πρέπει να την αποφύγουμε με κάθε κόστος και δεν είμαι σίγουρος πως ε, αυτό το έχουμε σκεφτεί. Το θέμα της γλώσσας επίσης που χρησιμοποιείται όσον αφορά και τις ιδιαιτερότητες της ασφαλιστικής ε, αγοράς είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που πρέπει να διατηρηθούν σε ένα τυποποιημένο πλαίσιο. Ξέρω πως χρησιμοποίησα ήδη τέσσερα ε, λεπτά και με την αδειά σας θα ήθελα τα υπόλοιπα έξι λεπτά να τα χρησιμοποιήσω αργότερα. Μάλιστα. Θα το, θα λάβουμε υπόψη αργότερα, γιατί νομίζω πως Έχουμε, έχουμε την αίθουσα μέχρι τις 12.30 ε, η διερμηνία. Τι θα κάνω λοιπόν. Θα ακούσουμε τώρα τους βουλευτές, αλλά δεδομένου το ότι αυτή τη στιγμή εστιάζουμε στο έγγραφο βασικών πληροφοριών, αν θέλουν και οι άλλοι ε, δύο εμπειρογνώμες να σχολιάσουν, ευχαριστώ. Αλλά να ακούσουμε πρώτα απ' όλα τις εντεράσεις των βουλευτών που ίσως θέλουν να παρεμούν. Ο κύριος Χατζημαρκάκης πρώτος. και πάλι προσφώτω τον κύριο Μπουσόλο, ο οποίο ε, είναι σκιώδη ηγητή. Ο κύριο Μπουσόλο στηρίζει την ιδέα μια ενιαία προσέγγιση ε, ε, στο έγγραφο με τις βασικές πληροφορίες, το οποίο θα δίνεται στους μικροεπενδυτές σε ολόκληρη την Ένωση. Και συμφωνεί με τον κύριο για μια ενιαία προσέγγιση. Το άρθρο 6 έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι κρίσιμη σημασία οι μικροεπενδυτέ να αντιλαμβάνονται τι πληροφορίε που του δίνονται. Το έγγραφο βασικών πληροφοριών θα πρέπει να είναι σαφέ, ακριβέ και μη παραπλανητικό. Επίση, ο κ. Μπεζόλ συμφωνεί με τον εισηγητή στο ότι δεν θα πρέπει να περιέχει διαφημιστικές και πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός από οποιοδήποτε άλλο διαφημιστικό υλικό. Η διατύπωση όμως θα πρέπει να προσαρμοστεί γιατί υπάρχει εδώ πέρα επικάλυψη μεταξύ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 2α του κυρίου Παντσέρη. Ο κ. Ζωή έχει κάποιε επιφυλάξει για την τροπολογία 10 που αφορά τη γλώσσα στο μέρος του κράτους μέλους όπου πωλείται το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τα προϊόντα που αγοράζονται στο ίντερνετ. Εάν γαλλόφωνος αγοράσει κάτι στο διαδίκτυο από μια φλαμανδική τράπεζα, ε, αναμένει πως θα βρει το έγγραφο και στα ε, γαλλικά, γιατί ε, θα είναι στο Βέλγιο. Αυτό μπορεί να προκύψει συχνά καθώς υπάρχουν τώρα όλο και περισσότερε τράπεζε online. Οπότε η πρόταση αυτή μπορεί να είναι αντιπαραγωγική σε αντίθεση με την πρόθεση η οποία είναι σωστή όσον αφορά το περιεχόμενο του βασικού ε, εγγράφου και ζωή χρειάζεται πω κάτι πρέπει να γίνει για να βελτιωθούν οι διατάξει του άρθρου 8. Οι κίνδυνοι αναφέρονται πάνω από ένα σημείο και μπορεί να βελτιωθεί νομίζω το κείμενο όσον αφορά το κόστο. Θα πρέπει να αναφέρεται και το πιο σημαντικό να αναφέρεται κατά τρόπον ώστε να είναι ε, κατανοητή από τον επενδυτή. Αν κάποιος π.χ. αγοράζει κομμάτι επενδυτικού ταμείου, μπορούν να υπάρξουν πολλές προμήθειες, αλλά δεν αντιλαμβάνεται ο πελάτης τι είναι όλα αυτά ή εάν ισχύουν στην περίπτωσή του. Επίσης μπορεί να είναι χρήσιμο για τον μικροεπενδυτή να έχει πληροφορίες για το φορολογικό καθεστώς που ισχύει για αυτό το προϊόν στην χώρα όπου πωλείται. Ο σχεδόν εισηγητή επίση υποστηρίζει τον εισηγητή όσον αφορά το ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι απαιτήσει πληροφοριών όσον αφορά την απόδοση του προϊόντος. Επίσης πρέπει να επισημάνουμε το ότι οι παρελθούσε ε, αποδόσει δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικέ. Τέλος, ο κύριος Μπουσόη ε, θεωρεί πως ε, θα πρέπει να γίνει κάτι όσον αφορά την αποζημίωση ε, για τυχόν απώλειες. Ε, κάτι το οποίο συνδέει η Κομισιόν στο έγγραφο βασικών πληροφοριών. Ο εισηγητής το διαγράφει αυτό στο άρθρο 19. Ε, κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο γιατί αν και δεν υπάρχει, ακόμα και αν δεν υπάρχει άμεση σχέση με την ποιότητα του εγγράφου θα μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ο ε, καταναλωτής, κάτι το οποίο βεβαίω θα είναι δυσανάλογο. Υπάρχουν και άλλα σημεία συζήτηση, αλλά νομίζω πως ε, έχουμε μια καλή αφετηρία. Μάλιστα, Σα ευχαριστώ κυρία Χάντσλικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκπροσωπώ εδώ την κυρία Πιετικάναν. Η ε, κυρία Πιετικάναν ευχαριστεί τον εισηγητή για την γνωμοδότησή του και για τις προσπάθειές του. Η νομοθετική πρόταση στόχο έχει την αύξηση της διαφάνειας και την ενημέρωση των μικροεπενδυτών με σύντομες, συγκρίσιμες και ε, εύληπτες πληροφορίες. Επίσης, η πρόταση είναι ένα απαραίτητο στοιχείο της καλύτερης προστασίας των καταναλωτών στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και συνδυάζεται με πολλές άλλες προτάσεις, όπως είναι η αναδιατύπωση για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση του ΣΟΣΕΚΑ και τη ΜΙΦΙΔ. Θέλουμε ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο που συμβάλλει στην καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. σκόπιμη είναι και νομική μορφή του κανονισμού, γιατί έτσι θα εξασφαλιστεί μια ομοιόμορφη εφαρμογή της σημαντικής αυτής νομοθεσίας. Η κυρία Πιετικάινεν θεωρεί ότι καλό θα ήταν να βελτιώσουμε κάπως την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα σημαντικό θέμα είναι η έννοια του κινδύνου και το προφίλ κινδύνου συγκεκριμένου ΠΡΙΠ. Πολύ σημαντικό θέμα. Η κυρία Πιετικάριν δεν έχει ακόμη πιστεί ότι είναι σωστή η μέθοδος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό. Γιατί η, ο υπολογισμό του κινδύνου και η παρουσίαση της καλύτερης επίδοσης δεν είναι ίσως η καλύτερη λύση. Και μπορεί το αποτέλεσμα αυτό να είναι παραπλανητικό. Γιατί έχουμε πορίσματα που δείχνουν ότι ε, επενδύσεις προηγούμενων, επιδόσεις προηγούμενων επενδύσεων δεν είναι ο, ο μοναδικός δείκτης για την αποδοτικότητα του συγκεκριμένου επενδυτικού ταμείου για το μέλλον. Αλλά και για τα ΠΡΙΠ, οι κίνδυνοι που αφορούν συγκεκριμένο προϊόν ε, δεν είναι ίδιοι. Οι κίνδυνοι είναι διαφορετικοί ανάλογα με το προϊόν. Αυτή η διαφοροποίηση θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στα έγγραφα με τις βασικές πληροφορίες. Ίσως θα μπορούσαμε στις βασικές πληροφορίες να περιλαμβάνουμε διάφορα σενάρια επιδόσεων, όπως προτείνει ο εισηγητής. Η κυρία Πιετικά είναι να κρίνει ότι καλό θα ήταν να επεξεργαστούμε περαιτέρω αυτή την πρόταση. Ας μην ξεχνούμε ότι ο απομόνος του κίνδυνος δεν είναι κάτι αρνητικό κατά ανάγκη. Γιατί όσο πιο μεγάλο είναι ο κίνδυνο, τόσο πιο μεγάλη είναι τα κέρδη. Τελικά η επένδυση είναι σωστή. Βέβαια, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο άνθρωπος που αναλαμβάνει τον κίνδυνο να αντιλαμβάνεται και τη φύση και την έκθεση του κινδύνου που αναλαμβάνει. Και μερικές φορές ε, ο επενδυτής έχει παραπληνηθεί Εξαιτία της μεγάλη περιπλοκότητα και τη αδιαφάνεια των επενδυτικών προϊόντων. Για να λαμβάνει λοιπόν μεγαλύτερο ε, κίνδυνο ο πελάτης θα πρέπει να είναι σαφώς ενημερωμένος και τεκμηριωμένος για το, για το εύρος του κινδύνου. Επίση, η κυρία Πιετικάινεν θα ήθελε να αναφερθεί και στις διαφορετικέ μορφές κινδύνου. Μερικέ φορέ ο κίνδυνος προέρχεται από την ε, περίπλοκη δομή του επενδυτικού ταμείου. Επίσης ε, το θέμα της, του πληθωρισμού και των επιδόσεων του ταμείου μπορεί να είναι χαμηλότερες από τον πληθωρισμό. Όλα αυτά θα πρέπει να αναφέρονται στο έγγραφα με τις βασικές πληροφορίες. Ε, και το διοικητικό κόστος και το κόστος διανομής θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ε, στις πληροφορίες για το κόστος. Βέβαια, τέτοιε πληροφορίες ε, δεν είναι σίγουρο ότι τις κατέχει ο εκδότης του προϊόντος. Αυτό το τμήμα του εγγράφου θα πρέπει να το συμπληρώνει ο διαμεσολαβητής. Η κυρία Πιετικάινεν έχει πολλές επιφυλάξεις σε σχέση με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή της νομοθεσίας, ώστε να καλύπτει όχι μόνο package products, αλλά και άλλα προϊόντα όπως είναι άμεσες αποταμιεύσεις, SARS και άλλοι που είναι πολύ διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα από τα πακεταρισμένα προϊόντα, αυτά τα προϊόντα του πακέτου επενδύσεων. Βέβαια, όλα αυτά θα τα εξετάσουμε και στα πλαίσια της αναθεώρησης της νομοθεσίας. Επιφυλάξεις έχει η κυρία σχετικά είναι σε ό,τι αφορά το κατά πόσο είναι πόσα το έγγραφο με τις βασικές πληροφορίες. Και κατά πόσο λεπτομεριακό, κατά πόσο θα πρέπει να είναι εξονυχιστικό το έγγραφο αυτό. Είναι πολύ διαφορετικά τα επενδυτικά προϊόντα και άρα η έννοια ενός το εγγράφου είναι συζητήσιμη για το ΒΕΠ, ιδιαίτερα δεν υπάρχει μια ευρύτατη επιλογή και πολύ διαφοροποιη... διαφοροποιημένα ταμεία με διαφορετικά προφίλ κινδύνου. Όλα αυτά τα σημεία η κυρία Πιετικάνεν θα τα επισημάνει και στις τροπολογίες που θα καταθέσει και προσβλέπει σε συνέχιση της συζήτηση με τον εισηγητή και τους και Ευχαριστώ. Thank you very um, uh, Ευχαριστώ κυρία Στάιλερ. Μία διευκρίνηση. Θα ήθελα να ζητήσω από το πάνελ ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα οποία συζητήθηκαν τώρα και στην οδηγία η οποία είχε περάσει μέχρι τώρα ε, και η οποία υποτίθεται ότι ισχύει. Τι πληροφορίες έχουμε από την εφαρμογή της οδηγίας αυτής. replicating what is being successful in one and not doing something in another. So I'm just asking that's a point of clarification. Thanks. No, I... Κοιτάξτε και εγώ νομίζω ότι τίθενται ορισμένα ερωτηματικά σχετικά με την εμβέλεια εφαρμογής αυτών των συγκεκριμένων προτάσεων. Ο κ. Παντζέβη διευκρίνησε ότι θα ήθελε να μην υπάρξει μείωση αλλά αύξηση της εμβέλειας εφαρμογής, του πεδίου εφαρμογής. Ο κ. Ταραμπέλα είναι ο τελευταίος ομιλητής από πλευρά των μελών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω καταρχάς την πρόταση που έγινε. Πράγματι και οι διευκρινήσεις των εμπειρογνωμόνων οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση. Έχει εξελιχθεί ε, ο κόσμος των προϊόντων αυτών. Παλαιότερα τα προϊόντα ήταν μετά από αίτημα του ιδίου του πελάτη, αλλά σε ορισμένες τράπεζες σήμερα, έτσι όπως εφαρμόζεται και από ορισμένου ενδιαμέσους τραπεζών, ε, πηγαίνουμε περισσότερο θα έλεγα σε κάποια προϊόντα τα οποία κατά περίπτωση προσφέρουν στην τράπεζα μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους. Απαιτείται περισσότερη διευκρίνηση βέβαια των προϊόντων. Εγώ ήμουνα υπεύθυνο γνωμοδότηση για την ετικετοθεσία των προσυσκευασμένων προϊόντων. Ξέρω ότι πολλές πληροφορίες μερικές φορές λειτουργούν αρνητικά είτε σε υπολογιστή είτε πρέπει να διαβάζετε δύο-τρεις σελίδες ε, τις οποίες θα πρέπει να δεχθείτε ή να μην δεχθείτε στο τέλος της ανάγνωσης, ε, τις δέχεστε χωρίς να τις διαβάσετε συνήθως. Είναι δύσκολες οι πληροφορίες αυτές, ε, αλλά πλούσιες και γι' αυτό απαιτείται να υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα των πληροφοριών, το κόστος εξόδου, το επίπεδο κινδύνου, το θέμα της φορολογίας, Πρέπει να ξέρετε πώς φορολογείται το προϊόν, εάν ισχύει και με ποιο τρόπο ισχύει. Εν πάση περιπτώσει απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια. Αυτό είναι το βασικό. Διαφάνεια και γνώση από πλευράς του πελάτη των συνθήκων λειτουργίας του προϊόντος. Μιλήσαμε για την απόδοση μέχρι τη στιγμή ε, της επαναγοράς αυτό δεν μπορεί να είναι τμήμα της διαφήμισης γιατί αν πιστεύετε ότι πρέπει να αγοράσετε βλέποντας το τι συνέβη το προηγούμενο έτος αγοράζετε ακριβά και υφίσταστε τις συνέπειες το επόμενο. Παρ' όλα αυτά είναι ένα στοιχείο πληροφόρησης το τι έχει αποδώσει μέχρι τώρα ένα τέτοιο προϊόν. Απαιτείται λοιπόν να υπάρχει ένα σύστημα ενημέρωσης το οποίο να επιτρέπει τις συγκρίσεις Ξέρετε στα προϊόντα, τα στρόφιμα έχετε, τις θερμίδες, τα ζάχαρα, τις πρωτεΐνες, κάποια βασικά στοιχεία. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα έτσι ώστε να είναι ενήμερος ο πολίτης ο οποίος θέλει να επενδύσει. Σε κάθε τύπου θα έλεγα επένδυση και τοποθέτηση χρημάτων στο μέλλον μια τέτοια ρύθμιση είναι απαραίτητη. Καλώς κάποιος άλλος θα ήθελε το λόγο, όχι. θα επανέλθω στους δύο μιλητές εμπειρογνώμονες αλλά και οι υπόλοιποι δύο έχουν την δυνατότητα να πάρουν το λόγο αν το επιθυμούν. Ας μιλήσουμε με τους κύριους ομιλητές και μετά θα σας δώσω το λόγο πάλι. Ο κύριος Μπιερνό. Ευχαριστώ. Χαίρομαι για τα σχόλια που άκουσα γιατί πραγματικά δείχνουν μια ευαισθησία για τις ανάγκες του καταναλωτή. Σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο, αλλά δεν θέλουμε ένα έγγραφο με βασικές πληροφορίες που θα είναι ταυτόσιμο για όλα τα προϊόντα. Σε καμία περίπτωση. Οι ε, αρμόδιες εποπτικές αρχές, οι ευρωπαϊκές αρχές χρηματοπιστωτικής ε, εποπτείας, είναι σε θέση να προσαρμόσουν το έγγραφο σε κάθε περίπτωση ανάλογα με το είδος του επενδυτικού προϊόντος. Δεν είναι το ίδιο μία κατάθεση ή μία μετοχή ή μία δέσμη επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές, ένα πρίπ δηλαδή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την οδηγία για το σύντομο προσπέκτους, η επενδυτέ που καλούνται να λάβουν μια απόφαση σπάνια έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν εμπεριστατωμένα ένα μακροσκελές έγγραφο. Παρόλο που το προσπέκτο αυτό δεν είναι πολύ ογκώδες, πολλές φορές δεν είναι καν στη γλώσσα του επενδυτή. Γι' αυτό και το έγγραφο με τις βασικές πληροφορίες δίνει μια πολύ πιο κατάλληλη λύση και είναι ένα καλύτερο εφόδιο για τον επενδυτή που μπορεί πια πιο τεκμηριωμένα να λάβει την απόφασή του. Γιατί στο έγγραφο με τις βασικές πληροφορίες πραγματικά ε, εστιάζει την προσοχή του επενδυτή στι βασικέ ε, αποφάσει και στα θέματα που τον ενδιαφέρουν περισσότερο από ότι το προσπέκτο που είναι πιο μακροσκελές. Θα μπορούσατε να σχολιάσετε το θέμα του πεδίου εφαρμογή, Συμφωνείτε με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή. και επίση το δικαίωμα που είναι διαφοροποιημένο ανάλογα με το είδο του επενδυτικού προϊόντος. Δηλαδή, η δομή τη πληροφορίας θα πρέπει να σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος. Τι γνώμη έχετε για αυτές τις διαφοροποίησεις. Αν κατάλαβα καλά την ερώτηση, και εμεί είμαστε υπέρ τη επέκτασης του πεδίου εφαρμογή. Είμαστε υπέρ τη διεύρυνση αυτή. Θεωρούμε ότι κάθε κατάθεση, κάθε επένδυση ουσιαστικά αναβάλει τα έξοδα. Δεν αγοράζει κανείς σήμερα ε, ένα προϊόν, κάνει οικονομίες σήμερα, αποταμιεύει και επενδύει για να ε, καρποθεί αυτά τα προϊόντα αργότερα, τη στιγμή της, μετά, όταν βγει στη σύνταξη. Και όλα αυτά τα αποταμιευτικά προϊόντα, τα επενδυτικά προϊόντα, αυτή την ανάγκη προσπαθούν να ικανοποιήσουν. Χρειάζονται λοιπόν οι πληροφορίες αυτές, αλλά είναι απαραίτητες οι πληροφορίες και για τις ε, επαγγελματικέ συντάξει, για παράδειγμα γιατί ο καταναλωτής θα πρέπει να ξέρει περί τίνος πρόκειται για να μην εκτεθεί σε υπερβολικούς κινδύνους και να διαφοροποιήσει το επενδυτικό του πακέτο. Χρειάζεται λοιπόν σαφείς πληροφορίες για τι επαγγελματική σύνταξη δικαιούται, για παράδειγμα. Σε μερικές χώρες αυτό είναι απλό. Υπάρχει μία ασφαλιστική εταιρεία, αλλά σε άλλες χώρες ο εργοδότης έχει με ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών για τις επαγγελματικές συντάξεις. Γι' αυτό χρειάζεται έγγραφα με βασικές πληροφορίες και για τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάρτη. Καταρχήν, το παιδί εφαρμογή θα πρέπει να είναι όσο πιο ευρύ γίνεται. Και αυτή είναι η ιδέα των PRIPS, τη δέσμη επενδυτικών προϊόντων. Να έχουμε μια ομοιόμορφη και συνεπή προσέγγιση για να μην υπάρχουν επενδυτικά προϊόντα που εξαιρούνται. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, τις επαγγελματικέ συντάξεις, όντως ε, οι συντάξεις έχουν σημαντικές ιδιαιτερότητες και η συμπερίληψή τους ε, στα έγγραφα με βασικές πληροφορίες θα δημιουργήσει περιπλοκές. Αλλά πιστεύω ότι η αρχή των εγγράφων με βασικές πληροφορίες θα μπορεί να επεκταθεί και στις συντάξεις. Μερικές ε, ασφάλειες ζωής μιλούν για εγγύηση κεφαλαίου πέραν της πάγιας επιστροφής και του μεταβλητού σημείου επιστροφής. Οπότε κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε να το διεκδικήσουμε για όλα τα προϊόντα. Βέβαια, έτσι κινδυνεύουμε να έχουμε μια περιόριστη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή και πού θα βάλουμε την οριοθετική γραμμή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα ανέβρεση της ισορροπίας για κάποια ασφαλιστικά προϊόντα, δηλαδή επέκταση, εφόσον προσφέρουν κάποιες εγγύησεις. Από αυτήν την άποψη νομίζω ότι η πρόταση είναι καλή όσο έχει. Ε, ε, ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Ξεκινήσω λέγοντας πως ε, στηρίζουμε οπωσδήποτε την εισαγωγή ενός απλού εγγράφου το οποίο επιτρέπει στους πελάτες να συγκρίνουν και να καταλαβαίνουν εναλλάξιμα επενδυτικά προϊόντα. Αλλά πρέπει να δούμε λίγο το πεδίο εφαρμογής, γιατί υπάρχει εδώ πέρα μια γενή σύγκρουση μεταξύ διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής και της ευκολίας με την οποία μετά μπορεί να παραχθεί ένα τέτοιο τυποποιημένο έγγραφο. Όσο πιο ε, στενό το πεδίο εφαρμογής, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να έχουμε συγκρίσιμα εγγραφά. Εάν μετά μιλάμε για οποιοδήποτε επενδυτικό προϊόν, μετά δεν συγκρίνουμε ίδια πράγματα, αλλά συγκρίνουμε μήλα με αχλάδια κτλ. Και θα είναι βεβαίως η τυποποίηση μετά μεγαλύτερη πρόκληση. Και έτσι ερχόμαστε στο ερώτημα της κυρία Στάιλερ, δηλαδή τι μπορούμε να μάθουμε από το, τα ΟΣΕΚΑ τα ΟΣΕΚΑ είναι ε, προϊόντα ομοιογενή και καθορίζονται επακριβώς. Βεβαίω δεν είμαι ειδικό στο έγγραφο βασικών πληροφοριών των ΟΣΕΚΑ, αλλά ξέρω πως είχε προκλήσεις. Και μιλάμε για προϊόντα τα οποία είναι αυστηρά καθορισμένα και ομοιογενή. Οπότε πρέπει εδώ πέρα να είμαστε κάπως προσεκτικοί όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή. Γενικότερα για τα πρίψη. Νομίζω πως υπάρχουν επίσης προκλήσεις για το πώς θα έχουμε την ισορροπία μεταξύ ενός σύντομου εγγράφου με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχει κατά την πώληση ο πελάτης και αν θεωρούμε πως όλα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με ένα σύντομο έγγραφο πρέπει να δούμε πως μπορούμε να ειδοποιήσουμε τους πελάτες για το που μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και επίσης αυτό σχετίζεται με ε, προϊόντα τα οποία έχουν πολλές επιλογές ταμείων μέχρι και εκατοντάδες ε, κατά μία. και είναι δύσκολο μετά να έχουμε ένα τυποποιημένο έγγραφο. Επίσης υπάρχει και η πρόκληση βεβαίως του ε, της ατομικής ε, επιλογής γιατί ειδικά για τα ασφαλιστικά προϊόντα υπάρχουν πτυχές του προϊόντος ε, το ασφάλιστρο, το κόστος που καθορίζονται από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του πελάτη και πάλι εδώ πέρα υπάρχει η πρόκληση για ένα ενιαίο τυποποιημένο έγγραφο το οποίο θα αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη Ευχαριστώ πολύ εγώ θα συμφωνήσω ίσως σας προξενήσει έκπληξη με κάποια από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Όξλη. Πράγματι, όταν το βλέπει κανείς και από αμυγός ασφαλιστικής πλευράς, αυτό που βλέπει κανείς είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο συντάσσεται η πρόταση σήμερα δεν δίνει την δυνατότητα να εκφραστούν σωστά τα ειδικά χαρακτηριστικά της ασφάλισης. Ο τρόπος με τον οποίο ε, περιγράφεται το κάθε προϊόν ε, αφορά αποκλειστικά το συγκεκριμένο προϊόν. Είναι κάτι όμως το οποίο θα πρέπει εν μέρη να παραμείνει και στις, επι, επι, στις μελλοντικές ρυθμίσεις. Σχετικά, όταν έχει κανείς ένα ασφαλιστικό προϊόν, έχει και ένα στοιχείο κάλυψης κινδύνου και υπάρχει και η δυνατότητα μερικές φορές να μην υπάρξει η δυνατότητα απόδειξης του συγκεκριμένου κινδύνου και για τις εγγυήσεις το ίδιο. Δεν υπάρχει τρόπος απόδειξης μιας τέτοιας εγγύησης η οποία να στηρίζεται, να εδράζεται σε, ε, σε συγκεκριμένα κεφάλαια. Όσο ευρύτερα κανείς λοιπόν θέλει ε, να υπάρξει η εφαρμογή, τόσο περισσότερες προκλήσεις θα δημιουργηθούν σε σχέση με την δυνατότητα ε, του να μπορεί να κάνει κανείς μια αποτελεσματική σύγκριση ανάμεσα στα διαφορετικού τύπου προϊόντα. Πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και θα πρέπει επίσης να δούμε τι θα κάνουμε και με τα προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν υψηλούς κινδύνους, αλλά πέραν αυτών ίσως θα είναι μια υπερβολή και είναι κάτι το οποίο θα καταστήσει τη σύγκριση ανάμεσα σε ανομοιογενή προϊόντα δύσκολη. Τώρα, για την ενημέρωση, στόχος μας θα είναι να ενημερώσουμε καλύτερα και όχι περισσότερο. Όταν βλέπει κανείς την ισχύουσα κατάσταση, διαπιστώνει κανείς ότι ένας ενδιάμεσος πουλά ένα προϊόν ασφαλιστικό, ένα προϊόν ζωής και πρέπει να δώσει πληροφορίες για 49 διαφορετικά πεδία προκαταρκτικά. Όταν βλέπει κανείς ε, ε, σχετικά με τα ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να δώσει ενημερώσεις για 70 στοιχεία επιπλέον. Um, Εάν πράγματι θέλει κάποιος να συγκρίνει αποτελεσματικά ορισμένα προϊόντα και αυτό το έχει αποδείξει και η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαιτείται μεγαλύτερη στοχοθέτηση, καλύτερη συγγνώμη στοχοθέτηση. Ε, σε ένα ασφαλιστικό προϊόν ο καταναλωτής ενδιαφέρεται όχι μόνο ε, για το τίμημα αλλά και για το πεδίο των καλυπτωμένων κινδύνων. Και γι' αυτό παρακαλώ δεν θα πρέπει να διευρύνουμε υπερβολικά το πεδίο εφαρμογής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Σας ευχαριστώ θερμά. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κύριε Παντζέρη, μήπως θέλετε λίγα σύντομα τελικά σχόλια και να επιβεβαιώσουμε και το χρονοδιάγραμμα για την επόμενη συζήτηση και μετά να δώσω το λόγο στην κυρία Στάιλερ για να μας μιλήσει για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Ο κύριος Παντζέρη. Πάρα πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Ο χαρακτήρας της συζήτησης κατέστησε εφικτή την ανταλλαγή απόψεων με τους τέσσερις εμπειρογνώμονες και σε σχέση με το στοιχείο του πεδίου εφαρμογής, ε, ιδιαίτερα για τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όχι τόσο όμως για τα ασφαλιστικά. Εμένα πάντως δεν μου φαίνεται να υπάρχουν ε, ασυμβατότητες ε, με την ε, οδηγία προοπτικών. Με την οδηγία τη λεγόμενη προσπέκτους καλύτερα. Θα πρέπει να προσπεθήσουμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο στόχος προς τον οποίο οδεύουμε. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε μία πορεία ξεκάθαρη ένα δίκτυο ξεκάθαρο το οποίο θα κρατά ενήμερο και θα ενημερώνει συστηματικά και συνεχώς τον πελάτη και για άμεσες και για έμεσες μορφές επένδυσης. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε διαφοροποιημένα προϊόντα, αλλά και σε παρόμοια προϊόντα θα πρέπει η ενημέρωση να είναι ενιοποιημένη, ενιαίας μορφής. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν αξεπέραστα προβλήματα αν να λύσουμε την κατάσταση στε βάθος. Τώρα για το γλωσσικό. Θα πρέπει να βρούμε μια καλύτερη έκφραση ιδιαίτερα για τα προϊόντα τα οποία αγοράζει κανείς διαδικτυακά. Και θα πρέπει επίσης να περιγράφονται σωστά τα κόστη στο προϊόν το οποίο προτείνεται διαδικτυακά προς τον καταναλωτή. Τέλος, θα πρέπει επίσης να βρούμε μια σωστή λύση και για τους ενδιαμέσους. Έχουν μια αντικειμενική ευθύνη, δεν είναι ξένοι στη διαδικασία της ενημέρωσης, παίζουν κεντρικό ρόλο για την παροχή της ενημέρωσης, για τα προϊόντα τα οποία προτείνει στον καταναλωτή έτσι ώστε να κάνει την τελική επιλογή. Ευχαριστώ λοιπόν τους σκιώδεις εισηγητές για τη συζήτηση που προηγήθηκε. Είμαστε στην αρχή ακόμα ή εν πορεία καλύτερα και ελπίζω να καταλήξουμε σε μια λύση η οποία να καλύπτει τις ανάγκες του καταναλωτή. Ευχαριστώ πολύ. Μην ξεχνάτε το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε το σχέδιο γνωμοδότηση. Η διορία για την κατάθεση των τροπολογιών λήγει στις 28 Ιανουαρίου. Εξέταση τροπολογιών στις 21 Φεβρουαρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή 4 Μαρτίου, γιατί η κατ' ουσίαν αρμόδια Επιτροπή θα ψηφίσει στις 26 Μαρτίου, γι' αυτό προσπαθήσαμε να επιταχύρουμε και το δικό μας χρονοδιάγραμμα. Αλλά ήταν πολύ χρήσιμη, νομίζω, η συμμετοχή και των εμπειρογνωμόνων στη φάση αυτή και χαίρομαι που τα καταφέραμε να το διοργανώσουμε. Ας περάσουμε τώρα στην επόμενη συζήτηση την αναδιατύπωση της, ασφαλισ... οδηγίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Η κυρία Στάιλερ είναι η συγκεκριά μας, έχει καταθέσει το σχέδιο γνωμοδότησής της. Ακούσαμε ήδη στον πρώτο γύρο τους καλεσμένους μας. Αλλά να πω και για τον κόσμο που μας παρακολουθεί από το διαδίκτυο. Θα ακούσουμε πρώτα τον κύριο Όξιλη, που είναι αρμόδιος για την πολιτική της οδηγίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών. Είναι επαΐων στα θέματα αυτά. ακούσαμε την κυρία Κόλλαρ που είναι Γενική Διευθύντρια της Insurance Europe που είναι Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εταιριών και ασχολείται ιδιαίτερα εδώ και πολλά χρόνια με το θέμα των ασφαλίσεων στις Βρυξέλλες. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία τις απόψεις τους και την παρουσίασή τους. Και μετά θα δώσω και πάλι το λόγο στους κύριους Κάρτη και Μπιερνιό πριν γίνει η συζήτηση και με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Έχουμε τρία τέταρτα, δεν είναι και πολλή ώρα, αλλά αν οι εμπειρογνώμονές μας περιοριστούν στο δεκάλεπτο, θα τα καταφέρουμε. Πρώτα όμως θα δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μα, την κυρία Στάιλερ, για τα εισαγωγικά σχόλια, για την παρουσίαση της γνωμοδότησής της πρώτα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που ξεκαθαρίσατε πως όλοι οι ομιλητές θα, μιλήσουν γιατί νομίζω πως έχουν άποψη και για την ε, ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Νομίζω πως έχουμε λοιπόν εδώ πέρα μια καλή αφετηρία. Η πρώτη πρόταση επέτυχε πάρα πολλές αλλαγές για την προστασία των σημερών των καταναλωτών. Ξέρουμε πως η οικονομική κρίση ε, μια ανάγκη για καλύτερη προστασία των καταναλωτών για μη παραπλαντικές πωλήσει και βελτίωση των ε, πρακτικών πώληση. Η αρμοδιότητά μας, όπως είπα, είναι ακόμα αντικείμενο συζήτησης. Ελπίζω να ασχοληθούμε με την προστασία των καταναλωτών και στις δύο επιτροπές. Έχουμε λοιπόν τους ομιλητές και λίγο χρόνο. Θα ε, είμαι λοιπόν σύντομη για την ε, έκθεσή μου. Το πεδίο εφαρμογής έχει επεκταθεί έτσι ώστε να καλύπτει και τα site σύγκρισης ε, τιμών, ίσως στην ίδια κατηγορία με τους, ενδιάμεσους, με τους ενδιάμεσους και θα καθορίσουμε επίσης αυτή την κατηγορία αντί να την ε, κατονομάζουμε απλώς για να μην βρεθούν παραθυράκια. Επίσης όσον αφορά την ε, δέσμευση διαφόρων προϊόντων έχω προτείνει την απαγόρευσή τους γιατί δεν υπάρχει αρκετό όφελος για τους καταναλωτές. Επίσης τα προϊόντα τα οποία θέλουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να μπορέσουμε να τα προστατεύσουμε όσον αφορά την υποχρεωτική ε, αμοιβή και την ε, υποχρεωτική επίσης αποκάλυψη ε, θεωρούμε πως εδώ πέρα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό κίνητρο για την σωστή ενημέρωση των πελτών επίσης θα πρέπει να δούμε και το ζήτημα των στόχων και της καλύτερης εξυπηρέτησης ε, των ε, συμφερόντων του πελάτη. Επίσης θα πρέπει αντί να χρειαστεί να το ζητήσει ο πελάτης ε, τα τυχόν συμφέροντα να αποκαλύπτονται είτε υποχρεωτικά είτε κατόπιν είτε προαιρετικά επίσης. Για το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογή θα πρέπει οι εγγεγραμμένοι ενδιάμεση εντό Ένωση να μπορούν να συνεργάζονται με αυτού εκτό Ένωση και να υπάρχει νομική σαφήνεια. Τέλος, το άρθρο 14 για την προσφυγή θα πρέπει ε, να διασφαλίσει μια συνοχή με τις υπόλοιπες οδηγίες. Επίσης, όσον αφορά τις ε, πράξεις ε, κατεξοδότηση και τη συνοχή, όπως είπαμε, την οδηγία MIFID 2, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ελάχιστη εναρμόνιση, γιατί αν οδηγηθούμε σε πάρα πολλές πράξεις εξουσιοδότηση θα δημιουργηθεί νομική αβεβαιότητα και για τον κλάδο και για τον καταναλωτή. Αναμένω λοιπόν τις τροπολογίες των συναδέλφων και την συνεργασία με τους κοιόδης και στην Επιτροπή Οικονομικών για να έχουμε μια οδηγία η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των καταναλωτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την εισαγωγή αυτή και για την δουλειά που έχετε κάνει στην έκθεση αυτή. Τώρα λοιπόν θα ζητήσω από τον κύριο Όξλεϊ να ξεκινήσει την ε, συζήτηση. Για 10 λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επιτροπή που μας δίνει ευκαιρία να μιλήσουμε για την δεύτερη οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Να ξεκινήσω λέγοντας πως η αρχή χρηματαγορών του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πάρα πολύ θετική για την δεύτερη αυτή οδηγία, καθώς έτσι επεκτείνεται η οδηγία και σε άλλες οντότητες οι οποίες πουλάνε ασφάλειες. Επίσης, ε, ιδιαίτερα χαιρόμαστε για το ότι και ασφαλιστικές επιχειρήσεις καλύπτονται. Νομίζω πως έτσι εδώ πέρα έχουμε ίση μεταχείριση για την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων. Χαιρόμαστε επίσης για το ότι υπάρχει εδώ πέρα αυξημένο επίπεδο ασφαλείας για τα ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα και μεγαλύτερος ρυθμιστικός έλεγχος, δηλαδή οι νέες διαδικασίες καταγραφής των ενδιαμέσων και οι πολύ αυστηρότερες διαδικασίες για διασυνοριακές δραστηριότητες είναι κάτι το θετικό. Όμως υπάρχουν ε, προβληματικοί τομείς και ίσως είναι χρησιμότερο για μένα να εστιαστώ σε αυτούς. Θα ξεκινήσω ε, από τα ε, αντικρώμενα συμφέροντα και την ε, αποκάλυψή τους. Επί της αρχής καλωσορίζουμε την πρόταση της Κομισιόν να απαιτεί την παροχή πληροφοριών στους πελάτες στο σημείο πώλησης για τις υπηρεσίες που παρέχει η ασφαλιστική εταιρεία. Πρέπει δηλαδή να λένε στους πελάτες με ποιον έχουν να κάνουν, για ποιο, ποιανού το λογαριασμό δρά ο ασφαλιστής, είτε δηλαδή ε, είναι για την ασφαλιστική εταιρεία, είτε για τον πελάτη ή και για τους δύο. Και αν το πρόσωπο αυτό τους δίνει κάποια συμβουλή και αν γίνεται αυτό ε, επί ποιας βάσης. Επίσης συμφωνούμε με την επιθυμία της Κομισιόν ε, για τα συχνά άσχημα αποτελέσματα προκύπτουν από τέτοιες πρακτικές. Αναγνωρίζουμε πως συγκρούσεις αυτές υπάρχουν, συγκρούσεις συμφερόντων και, για να τα πούμε απλά, ο τρόπος με τον οποίο πληρώνονται οι εταιρείε και τα άτομα εντός των εταιρείων μπορεί να οδηγήσει στο ποιες συμβουλές θα δοθούν ε, στους καταναλωτές για το σε ποια προϊόντα θα πρέπει να επενδύσουν. Και άρα εδώ πέρα υπάρχει ένα κίνδυνο, ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν είμαστε τόσο πεπισμένοι για το ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι η σωστή. Η Κομισιόν προτείνει ένα καθεστώς υπό το οποίο οι ενδιάμεσοι ασφαλιών ζωής θα πρέπει να δίνουν λεπτομέρειες για την αμοιβή τους στους πελάτες οι ενδιάμεση γενικών ασφαλιών θα δίνουν αυτή την πληροφορία κατόπιν αιτήματος και οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι ενδιάμεση θα πρέπει να δίνουν λεπτομέρειες για το επίπεδο αμοιβών των υπαλλήλων. Ενστικτοδός βεβαίως το να δίνονται περισσότερες πληροφορίες στους πελάτες φαίνεται καλή ιδέα. Ε, υπό ένα μοντέλο λογικού καταναλωτή κάποιος ο οποίος έχει περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει τις, ε, τα συγκρόμενα συμφέροντα που υπάρχουν πιθανώς εντός του ενδιάμεσου ή της ασφαλιστικής εταιρεία. Και έτσι θα μπορέσουν να κάνουν συγκρίσεις και να βρουν καλύτερα προϊόντα. Αυτό μετά βεβαίω θα οδηγήσει σε ανταγωνιστική πίεση της εταιρεία και στο να αλλάξει συμπεριφορά τους. Και η επιτυχία βεβαίως θα εξαρτηθεί από τι αγορές, από τον καταναλωτή, το προϊόν και από την ικανότητα του καταναλωτή να κινηθεί στην αγορά. Η εμπειρία μας είναι πως για μη επενδυτικούς ε, πελάτες ασφαλιών δεν συμβαίνει αυτό πάντα. Για να μπορέσει ε, να είναι αποτελεσματική η αποκάλυψη της αμοιβή πρέπει να μπορεί να αντιληφθεί τις πληροφορίες αυτές ο πελάτης και μετά πρέπει να αλλάξει τη συμπεριφορά του ε, με τρόπο ώστε να βγει σε καλύτερο αποτέλεσμα. Και η εμπειρία μας είναι πως αυτό δεν σημαίνει πάντα. Οι πελάτες δεν διαβάζουν πάντα τις πληροφορίες που τους δίνονται, όταν τις διαβάζουν δεν τις καταλαβαίνουν πάντα, ειδικά όταν υπάρχει ένα κίνητρο για τις εταιρείε να καταστήσουν ε, ακατανόητες αυτές τις πληροφορίες και αν τις καταλάβουν δεν τις απορροφούν πάντα και δεν τις χρησιμοποιούν για να συγκρίνουν με άλλες προσφορές. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και χειρότερα αποτελέσματα γιατί κολλάνε οι καταναλωτές στο επίπεδο της προμήθειας. Δηλαδή είναι ίδια τα ασφάλιστρα αλλά διαφορετικό το επίπεδο προμήθειας πάνε σε αυτό το οποίο έχει χαμηλότερη προμήθεια αλλά ίσως να μην είναι το καταλληλότερο προϊόν και βασικότερο η ε, αποκάλυψη του επίπεδου της αμοιβή δεν καλύπτει το ζήτημα των δεν καλύπτει ε, το ζήτημα της οργάνωσης ε, η οποία θα μπορούσε ίσως να αποτρέψει τέτοια αντικρώμενα συμφέροντα. Δηλαδή θα πρέπει να δουν οι εταιρείε που υπάρχουν αυτά τα αντικρώμενα συμφέροντα και να τα διαχειριστούν και να τα μειώσουν. Αυτή είναι η προσέγγιση που υπάρχει στην οδηγία MIFID. Δεν θεωρούμε πως οι πελάτες δεν θα πρέπει να έχουν πληροφορίες για τις αμοιβέ. Αν θεωρούν πως ε, χρειάζονται αυτές τις πληροφορίες και τις ζητήσουν, οπωσδήποτε πρέπει να τις έχουν. Αλλά να τις έχουν μαζί με μια διαδικασία διαχείρισης των ε, δικρόμενων συμφερόντων. Κάποια άλλα ε, ζητήματα στα τέσσερα λεπτά που μου απομένουν. Όπως είπα, εμείς είμαστε υπέρ των ε, αυστηρότερων προδιαγραφών πώληση για επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα. Αλλά θέλουμε μια σύνοχη για τις ε, εταιρείε ε, και στην οδηγία μη και στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Χρειάζεται μια ενιαία προστασία των καταναλωτών, είτε μιλάμε για ε, ένα καθαρά επενδυτικό προϊόν, είτε ένα επενδυτικό ασφαλιστικό προϊόν. Γιατί ο πελάτης δεν ενδιαφέρεται για την συμβατική βάση αυτού του προϊόντος. Χρειάζεται μια ενιαία προστασία. Κάτι για το πεδίο εφαρμογής. Όπως είπα, είμαστε υπέρ της επέκτασης του και σε άλλες εταιρείες που πουλάνε ασφάλειες, αλλά έχουμε ανησυχίες για την επέκταση σε εταιρείες οι οποίες ε, ε, κάνουν παραδείγματος χάρη την αξιολόγηση για τις αποζημιώσεις που οι ασφαλιστικές εταιρείες γιατί υπάρχει η ρυθμιστική ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρείας για τις εταιρείες ε, εμπειρογνωμόνων και αν επεκταθεί αυτό και σε εταιρείε εμπειρογνωμόνων ε, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε το απαραίτητο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Είμαστε υπέρ της βελτίωσης των επαγγελματικών προδιαγραφών αλλά όπως είπε και η κυρία Στάιλερ, ανησυχούμε για το ότι υπάρχουν πολλές πράξεις εξοδότηση στην πρόταση για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και θα θέλαμε να δούμε ένα ξεκάθαρο κείμενο και όχι την αβεβαιότητα που προκύπτει από τις πράξεις εξοδότηση. Επίσης, οι πολλαπλές πωλήσει ε, διαφορετικών προϊόντων ανισχούμε, δεν ξέρουμε. Θεωρούμε πως θα μπορούσαμε να έχουμε εδώ πέρα μια επιγράμμιση της ασφαλιστική ενσουλάσης με την οδηγία για τι αγορέ χρηματοπιστωτικών μέσων. Επίσης, για την εναλλακτική επίλυση διαφορών και την εξοδικαστική επίλυση διαφορών υπάρχουν κάποιοι όροι που επιβάλλονται στα κράτη-μέλη για την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Είναι κάτι το θετικό και οι εταιρείε θα πρέπει να υποχρεούνται να συμμετέχουν στην εναλλακτική επίλυση διαφορών, αλλά οι όροι ε, νομίζω θα διαβρώσουν την προστασία των καταναλωτών, ειδικά καθώς απαιτείται πως δεν θα είναι υποχρεωτικές οι αποβάσεις ε, για τις ε, εταιρείε. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε αρκετά χρήσιμα στοιχεία. θα υπάρξει ένα συνολικότερο πακέτο και μέσα στο πακέτο αυτό θα πρέπει να υπάρχει συνεχή στις προτάσεις. Η επόμενη ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ που προσκαλέσατε την Insurance Europe. Φυσικά και είμαστε υπέρ της βελτίωσης της προστασίας του καταναλωτή για όλες τις δυνατότητες αγοράς ασφαλιστικών προϊόντων. Αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε και τις απαιτούμενες πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να παρέχονται με σωστό τρόπο. Όλα τα μέτρα τα οποία προτείνονται με τους διάφορους τρόπους, IND και CRIPS, θα πρέπει ε, αποδεδειγμένα να προσφέρουν και να ωφελούν τον καταναλωτή. Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να θέσω τρεις στόχους. Πρώτον, θεωρούμε ότι η εξυπηρέτηση των στόχων αυτών δεν θα πρέπει να εξυπηρετήσει μόνο την βιομηχανία, την ασφαλιστική, αλλά και τους καταναλωτές. Αυτός είναι ένας βασικός στόχος. Έχει σημασία της διατήρησης επίσης της πολλαπλότητας των τρόπων, των διάβλων διάθεσης των προϊόντων. Έχουμε τις ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες διαθέτουν τα προϊόντα τους άμεσα, ε, μέσω των υπαλλήλων τους, μέσω του διαδικτύου. Έχουμε ένα ευρύτατο δίκτυο όπου ε, διαχέεται η ασφάλιση μέσω του πιστοτικού συστήματος. Έχουμε μερικής απασχόλησης ε, πράκτορες, υπαλλήλου, ενδιαμέσους. Όλα αυτά τα, όλοι αυτοί οι διάβλοι παρέχουν μια πολλαπλότητα επιλογών κρίσιμη για τον καταναλωτή και αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερα θετικό. Αυτό το οποίο ζητά ο κόσμος είναι να μην υπάρχουν διακρίσεις εις βάρος ή ασδήποτε από αυτές τις μορφές διάθεσης των ασφαλιστικών προϊόντων. Όλες αυτές οι δυνατότητες διάθεσης θα πρέπει βέβαια να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο το οποίο να είναι ισορροπημένο, αναλογικό και ωφέλιμο για τον καταναλωτή τελικά. Αυτό θα μας βοηθήσει να υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε αγορές μετά από συζήτηση και συμβουλές ή σε αγορές άμεσα μέσω διαδικτύου και κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα της ενημέρωσης για τους καταναλωτές. Είναι κάτι το οποίο σαφώς θα πρέπει να βελτιωθεί. Απαιτούνται καλύτερες πληροφορίες Εγώ και στην προηγούμενη παρέμβασή μου είπα ότι το περισσότερο είναι εχθρός του καλού. Νομίζω ότι η πείρα μέχρι τώρα δείχνει ότι λεπτομερείς εξηγήσει ε, είναι εις βάρος των καταναλωτών και πολλές φορές παραπλανούν τον καταναλωτή. Θα πρέπει επίσης να αποφύγουμε περιτές πληροφορίες και στα πλαίσια αυτά θα χρειαστεί να συνεχίσουμε και την συζήτηση σχετικά με την αποκάλυψη των αμοιβών, των αποδόσεων, τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Να δούμε αν η αμοιβή, σαν παράδειγμα των ενδιαμέσων, είναι καταποκοπήν ή είναι ποσοστιαία της απόδοσης ε, νομίζω ότι η πρόταση η οποία γίνεται είναι μια καλή, ισόρροπη πρόταση και μπορεί να ενημερώσει αρκετά σωστά τον καταναλωτή. Να πω επίσης ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον κατελάχιστον εναρμόνισης, ως εκ τούτου απαιτείται κατελάχιστον νομοθέτηση αλλά οι αγορές υπάρχουν. Οι αγορές και τα κράτη-μέλη μερικές φορές έχουν ξεπεράσει το επίπεδο στο οποίο εμείς στοχεύουμε και έχουν καταλήξει σε αυτό το οποίο θεωρούν σαν την καλύτερη δυνατή βάση. Πάντα σε επίπεδο ενημέρωσης θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να επανέλθω στα ειδικά χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού τομέα. Τα είπα αυτά και στην αρχική μου παρέμβαση. Να πω ότι σε αυτή τη φάση δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποδείξουμε ξεκάθαρα τα ειδικά χαρακτηριστικά της ασφάλισης. Πάντως οι οδηγίες αυτές πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να απομονωθούν μεταξύ τους. Εργαζόμαστε και στα πλαίσια της Solvency 2 και εκεί τίθεται το θέμα της ε, σωστής ενημέρωσης πριν από την υπογραφή των συμβάσεων και απαιτείται στη συγκεκριμένη περίπτωση να υπάρξει επικάλυψη στην ενημέρωση των καταναλωτών όπως επίσης και παραπλανητικές μορφές ενημέρωσης των καταναλωτών και στις ασφαλίσεις και στα υπόλοιπα προϊόντα. Έτσι θα διασφαλίσουμε την επιλογή των καταναλωτών. Θα πρέπει στο μέλλον οι καταναλωτές να είναι σε θέση να αγοράσουν ή οδήποτε ασφαλιστικό προϊόν με τον τρόπο τον οποίο επιθυμούν. Οι διαδικασίες θα πρέπει να απλοποιηθούν. Γνωρίζουμε βέβαια ότι πάρα πολλοί καταναλωτές δεν θέλουν συμβουλές, δεν θέλουν ενημέρωση ιδιαίτερα για ορισμένα πολύ απλά, μη περίπλοκα ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία υπάρχουν. Σαν παράδειγμα ασφάλεια για τα κατοικίδια ζώα ή ασφάλεια ε, για ε, την κατοικία των ε, ασφαλιζομένων, απλές μορφές ασφάλειας γενικότερα. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να αγοράζουν ένα τέτοιο προϊόν ακόμα και χωρίς να ενημερώνονται εφόσον αυτό επιθυμούν βέβαια σε ορισμένες ασφαλιστικές αγορές συζητείται επίσης ο καταναλωτής να πληρώνει την ενημέρωση την οποία θα ζητά από τον ασφαλιστή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, ε, πρέπει να τεθεί σε συζήτηση εφόσον κάποιες αγορές βέβαια το επιθυμούν. Τώρα για τη συνεκτικότητα των προτάσεων ανάμεσα στο AMD και στο MIFED Νομίζουμε ότι για τις διασταυρούμενες πωλήσει ε, ε, θα πρέπει να υπάρξει γράμμιση με την οδηγία MIFED και να μην υπάρχουν στρεβλώσεις ε, στον ανταγωνισμό. Υπάρχουν, εδώ είναι κάτι που μας ανησυχεί, υπάρχουν πάρα πολλές κατεξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες είναι δύσκολα ερμηνεύσιμες και εξηγήσιμες. Και τέλος, Δεν θα πρέπει να υπάρξει έλλειψη εμπιστοσύνης. Ε, μιλάμε για την διαιτησία στον τομέα των ασφαλιστικών προϊόντων και θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα ρύθμισης επίσης και των ζημιών και απολειών. Ευχαριστώ. Πολύ σαφή τα σχόλια. Θα επανέλθουμε σε αυτά. Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Κάρτη για να μας σχολιάσει τη δεύτερη πρόταση για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σχολιάσω καταρχήν τις εισαγωγικές παρατηρήσεις της κυρίας Στάιλερ. Συμφωνούμε ότι η δεύτερη οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι καλύτερη από την πρώτη οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Και μάλιστα μόλις που είχε στεγνώσει μελάνη τις πρώτες οδηγίες όταν αποφασίστηκε η αναδιατύπωση ε, με τη δεύτερη οδηγία, κάτι που είναι ιδιαίτερα δαπανηρό για τους διαμεσολαβητές. Παρόλο που αναγνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη η ενημέρωση της οδηγίας. Επίσης θα πρέπει να αποφευθούν τα παραθυράκια, να περιοριστούν όσο γίνεται ιδιαίτερα για τις ε, πωλήσει μέσω διαδικτύου. Επίσης για, τους, για τις μορφές προσαρμογής και αντιστάθμισης των δαπανών, των, απολυ... των ζημιών, συγγνώμη, και αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό και αφορά και το πεδίο εφαρμογή. Τώρα, σε ό,τι φορά την παροχή των πληροφοριών ε, για μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά που περιλαμβάνει πολλές μορφές διανομής και η διαμεσολάβηση είναι ο μεγαλύτερος τομέας, αλλά όχι ο μοναδικός τομέας διανομής. Αλλά ακόμη και ο όρος διαμεσολάβηση περιλαμβάνει πολλές κατηγορίες διαμεσολαβητών και μεσητών. Η πρωτορχική μας ανησυχία είναι να εξασφαλίσουμε ένα ευρύ φάσμα διαμεσολάβησης, ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για τον καταναλωτή και να αποφευθεί πάση θυσία η στρέβλωση του ανταγωνισμού ή η εύνοια ενός ε, μια ομάδας μόνο διαμεσολαβητών ει βάρο ε, των άλλων. Γιατί κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε κατακαιρματισμό τη αγορά, συρρήκνωσή τη και θα αποβεί εις βάρος του καταναλωτή. Επίσης, να δούμε και το θέμα τη δεύτερη οδηγία ασφαλιστική διαμεσολάβηση υπό το πρίσμα τη προστασία του καταναλωτή. Πρόκειται για ένα πακέτο και γενικώ το πακέτο αυτό είναι αρκετά ισορροπημένο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις, προδιαγραφέ ε, ε, τις προδιαγραφές, τα στάνταρ ε, μας προβληματίζει κάπως το θέμα των κατεξουδότηση πράξεων, αλλά οι αδρές γραμμές μας βρίσκουν σύμφωνος. Επίσης, κατάλληλες πληροφορίες στον καταναλωτή, στο σημείο πώλησης και ανασύμβαση, να αποφευθεί ε, ο φόρτος, ε, η πληθώρα των πληροφοριών, θα πρέπει να είναι αναλογικές. Επίσης, ε, το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Το ζήτημα αυτό, αν όχι άμεσα, έμεσα αναφέρθηκε και στην πρώτη οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Εδώ θα πρέπει να αναφέρεται ρητά και τα κατηγορηματικά και όχι μόνο έμεσα όπως στην πρώτη οδηγία. Επίσης θα πρέπει να εντοπίσουμε, να διαχειριστούμε και να μετριάσουμε τέτοιες συγκρούσεις συμφερόντων που μερικές φορές είναι εγγενείς ε, σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, το ίδιο και τις χρηματοπιστωτικές, αλλά θα πρέπει να διαχειριστούμε αυτές τις σύγκρουσεις συμφερόντων, να τις εντοπίσουμε πρώτα και να τις μετριάσουμε. Και φυσικά να επιστήσουμε την προσοχή του καταναλωτή σε αυτές στο σημείο της πώληση και πάλι περιπτωσιολογικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, η διαφάνεια σημαίνει εντοπισμό του διαμεσολαβητή, του πιο εκπροσωπεί, τις αποδοχές του, τις πηγές των αμοιβών. Όλα αυτά είναι στοιχεία της διαφάνειας. Επίσης θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στον καταναλωτή να ζητά λεπτομέρειες ως προς τις αποδοχές του διαμεσολαβητή όπως προβλέπει η παρούσα οδηγία, αλλά μόνο για μία πενταετία. Αλλά προσοχή, όπως είπα και στην αρχή, η αγορά αυτή είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική. Δεν θα πρέπει λοιπόν να απομονωθεί μία μόνο ομάδα ή να ευνοηθεί. Αλλιώς ε, με κάτι τέτοιο θα δημιουργηθεί στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αναφέρθηκε ε, θα πρέπει οι οδηγίες να είναι σχετικές, ε, αναλογικές υπάρχει διαφορά όμως μεταξύ των ασφαλιών ζωής και των ε, λοιπών ασφαλιών. Είναι πολύ διαφορετικά τα προϊόντα που πολλούνται σε μια ασφάλεια ζωής και στις λοιπές ασφάλειες. Τώρα, η αποκάλυψη πληροφοριών ε, ως προς τις αποδοχές σε λοιπές ασφάλειες εκτός ζωής, ε, οι υποχρεωτικές τέτοιες πληροφορίες μπορεί να έχουν τεράστιες συνέπειες. Και μία αφελής απλουστευμένη, απλοϊκή προσέγγιση υιοθετείται μερικές φορές και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει πραγματικά. Και εγώ διαμεσολαβητής είμαι και είμαι και πρόεδρος μιας ε, τέτοιας ε, εταιρεία. Ε, αλλά αυτή είναι η βασική μου δραστηριότητα. Και θα σας έλεγα ότι η αποδοχή μου είναι 20% η προμήθεια. Γνωρίζω όμως την αγορά μου ότι αν πάτε και ρωτήσετε μια τράπεζα ή κάποιον ασφαλιστή θα πει 20-21%, 22%. Ωραία. Αυτό που λέμε είναι το ποσοστό, αλλά αυτό που κρύπτουμε είναι ότι ο ασφαλιστής είναι που κάνει όλη τη δουλειά. Ενώ η τράπεζα ουσιαστικά δεν είναι σημείο αναφορά. Οπότε συγκρίνεται ανώμια πράγματα. Η αξία της αποδοχής για κάποιον θα μπορεί και 30%, αλλά ούτε και αυτό μας ενδιαφέρει θα πρέπει να δίνουμε την ευκαιρία στον καταναλωτή να θέτει την ερώτηση, αν θέλει οπωσδήποτε να μάθει, αλλά αν εγκαταστάσετε μόνο ένα διάβλο διαμεσολάβηση να αποκαλύψει τι πληροφορίες αυτέ, είναι σαν να προκαλείται στρέβλωση του ανταγωνισμού και συρρυκνώνεται το φάσμα επιλογών του καταναλωτή. Να επιλέξει τον κατάλληλο ε, ασφαλιστεί σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά. Και παραλαμβάνω διαφορά τεράστια μεταξύ ασφαλιών ζωής και λοιπόν ασφαλιών. Και μάλιστα εκεί έχουμε αιτήσια ανανέωση συμβάσεων και εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά. Γι' αυτό μια τέτοια υποχρέωση είναι κάπως επικίνδυνη. Ένα άλλο σημείο που με ενδιαφέρει ως διαμεσολαβητή είναι οι σχέσεις που έχω με τους πελάτες μου. Οι διαμεσολαβητές ενδιαφέρονται να έχουν διαβίου σχέσεις με τους πελάτες. Αυτό τους ενδιαφέρει. Να συνεχίσουν τη δραστηριότητά του, να μην χάσουν τους πελάτες τους. Και θέλουν κάθε χρόνο ανανέωση για δεκαετίες ολόκληρες. Αυτή είναι η αξία της ε, οικονομικής αυτής της δραστηριότητας. Δεν θέλουμε να πουλήσουμε μόνο μία φορά. Δεν έχουμε μία συνεχή και ε, συνεχώς ανα, ανα, ανανεώμενη σχέση με τον πελάτη. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας να είναι ευρύ, με ελάχιστες εξαιρέσεις και μόνο εφόσον δικαιολογούνται από έκτακτες και σπάνιες περιπτώσεις, οι πληροφορίες που να δίνονται στο πελάτη να είναι ε, και στη, στιγμή της πώληση, να είναι έγκαιρες, να είναι σχετικές με το αντικείμενο, όχι περιτές και υπερβολικές και μερικές από αυτές που προτείνει η Επιτροπή δεν έχουν αυτό το χαρακτήρα. Επίσης, ε, να γίνει διαχείριση της σύγκρουσης ε, συμφερόντων από την παροχή πληροφοριών προς τον πελάτη, ώστε ο πελάτης να αντιλαμβάνεται αν υπάρχουν κάποια κίνητρα ως προς τη συγκεκριμένη συμβουλή ή τις υπηρεσίες που του χορηγούνται στο σημείο της πώληση. Επαναλαμβάνω, βασικό μέλημα του κανονισμού είναι να εξασφαλιστούν συνθήκες ίσου ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων μορφών διαμεσολάβησης σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά. Γιατί αν αυτός ο στόχος δεν υλοποιηθεί, θα καταστραφούν ε, εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαμεσολάβησης που καθημερινά προσφέρουν τεράστιο έργο στην ευρωπαϊκή αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας άφησα να μιλήσετε λίγο περισσότερο γιατί εκτιμήσαμε την εμπειρογνωμοσύνη και το πάθος σας. Ο κύριος Μπέρνιο. Να αφήσουμε 10 λεπτά στην εισηγήτρια για να κλείσει το θέμα. Έχετε το λόγο κύριε Μπιερνό. Σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων, γιατί είναι το πιο θερμό θέμα σε αυτή τη φάση και μετά θα περάσω στο θέμα του πεδίου εφαρμογής. Σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων, συμφωνούμε με αυτά τα οποία είπε ο κ. Σόξλη, ότι δηλαδή η ενημέρωση δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση, δεν θεωρείται ότι καλύπτει τα προβλήματα που δημιουργούν οι συγκρούσεις συμφερόντων και τις τρευλώσεις που δημιουργούν στην αγορά. Καταρχάς το θέμα της αμοιβή του ενδιαμέσου. Ο ενδιάμεσος μπορεί να είναι μια μικρή επιχείρηση, μπορεί να είναι και μια τράπεζα. Η αμοιβή του ενδιαμέσου μπορεί να επηρεάσει κατά σημαντικό τρόπο την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Δεν μιλήσαμε αυτή τη στιγμή για τις λεγόμενες υποπροϋπόθεση αμοιβέ. Αυτό τι σημαίνει. Το επίπεδο της αμοιβή επηρεάζεται αν φτάσετε σε ένα συγκεκριμένο κύκλο εργασιών, όχι μόνο σε ένα προϊόν, αλλά σε ένα σφαιρικό λογαριασμό στη συγκεκριμένη επιχείρηση, τράπεζα, ασφάλεια κτλ. Έχετε λοιπόν την τάση να φέρετε όλα τα προϊόντα τα οποία διαχειρίζεστε σε μία επιχείρηση για να αυξήσετε τον κύκλο εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης και το χαρτοφυλάκιο του συγκεκριμένου πράκτορα ή ενδιαμέσου ακόμα και αν δεν είναι το καλύτερο για τον καταναλωτή. Και είναι φυσικά κάτι το αρνητικό για τις νέες επιχειρήσεις και τα νέα προϊόντα που θέλουν να μπουν στην αγορά. Θα δυσκολευτούν γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις συγκεντρώνουν τα πάντα. Μια άλλη μορφή υποπροϋπόθεση αμοιβή που γνωρίζουμε στο Βέλγιο είναι ότι η αμοιβή του ενδιαμέσου επηρεάζεται από το μέγεθος της βλάβης ή από τον αριθμό των ζημιών που έχει δηλωθεί από τον πελάτη. Αν είστε ένας ενδιάμεσος και αν πράγματι έχετε ένα πελάτη ο οποίος να έρχεται με μια αμφισβητούμενη ζημία, θα έχετε την τάση να του πείτε ότι δεν καλύπτεται η συγκεκριμένη ζημία για να μην επηρεάσετε τη δική σας αμοιβή από την επιχείρηση. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι εξαιρετικά κακή. Αυτά είναι παραδείγματα για να σας δείξω ότι θα πρέπει αυτές οι κα... υπό προϋπόθεση αμοιβέ να καταργηθούν γιατί είναι βλαβερές για τον καταναλωτή. Ένα άλλο θέμα είναι η αμοιβή των υπαλλήλων της τράπεζας, της επιχείρησης που λειτουργήσαν ενδιάμεσος ή υπάλληλοι ενός ενδιαμέσου μεσαίου μεγέθους ή μιας εταιρείας ασφαλιστικής. Τίποτα δεν ε, λέγεται πάνω στον τύπο και την οργάνωση των αμοιβών αυτών. Μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιεί όλα τα κίνητρα τα οποία θεωρεί απαραίτητα αν φτάσουμε ας πούμε σε ένα επίπεδο μιας γερμανικής εταιρείας η οποία προσφέρει σύντομες, σύντομα ταξιδάκια στην Βουδαπέστη για λίγες μέρες και μια γιορτή κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να φοράτε παπιγιόν και ένα μπρασλέ ενός ιδίου χρώματος είναι και αυτό ένα κίνητρο ε, για την επιδίωξη επίτευξης ε, στόχων, μερικές φορές αρνητικών για τον πελάτη. Σχετικά τώρα με τη διαφάνεια των ε, αμοιβών, ποιος πληρώνει την αμοιβή, ε, ο, ο καταναλωτής το κάνει αυτό. Είναι απαραίτητο λοιπόν, εφόσον δεν έχουν καταργηθεί όλες οι συγκρούσεις συμφερόντων, να υπάρχει πλήρης ενημέρωση. Και δεν μπορούμε να δεχτούμε μόνον ο καταναλωτής ο οποίος είναι σωστά ενημερωμένος ε, να προκαλεί την ενημέρωσή του. Γιατί συνήθως οι καταναλωτές αυτές πράγματι δεν έχουν και πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη ενημέρωση. Σχετικά τώρα με το πεδίο εφαρμογής, σύντομα. Η οδηγία ND1 εξαιρούσε τα ασφαλιστικά προϊόντα από την πώληση αγαθών, όπως σαν παράδειγμα ένα κινητό τηλέφωνο. Εξαιρούσε επίσης ε, ε, και τις ασφάλειες ε, ταξιδίων. Οι ασφάλειες τώρα ταξιδίων και ενοικίας της αυτοκινήτων εμπλέκονται στην οδηγία, περιλαμβάνονται αλλά με ένα ελαφρύ καθεστώς θα έλεγα. Και έρχομαι τώρα στην ασφάλιση αγαθών. Βλέπουμε σαν παράδειγμα ότι όλοι οι πολιτές όταν αγοράζετε το τηλέφωνο σας σας προτείνουν ε, ένα συμβόλαιο χωρίς να σας εξηγήσουν τις εξαιρέσεις και πληρώνετε αρκετά ακριβά και δεν γνωρίζετε ε, ε, ότι οι ενδιάμεσοι παίρνουν το 50% αυτού του ασφαλίστρου. Αγοράζεται ένα προϊόν ακριβό το οποίο μερικές φορές είναι και πάρα πολύ άχρηστο. Πρέπει λοιπόν στα πλαίσια της οδηγίας αυτής να υπάρξει μια κάποια αλλαγή με σωστή εφαρμογή των κανόνων συμπεριφοράς και ενημέρωσης των καταναλωτών και για τις ασφάλειες για τα τηλέφωνα και για τις ασφάλειες για ταξίδια όπου δεν σας εξηγούν πολλές φορές τις εξαιρέσεις, σαν παράδειγμα λόγω προβλημάτων υγείας. Ε, ενώ η ενημέρωση για όλες τις ασφάλειες θα πρέπει να είναι κάποιο επίπεδο και να δίδεται από τους ασφαλιστές και από τους ενδιαμέσους. Και μάλιστα αν κάτι τέτοιο μείνει εκτός της ε, οδηγίας ΜΙΦΕΔ, μένει και εκτός της οδηγίας για την προστασία του καταναλωτή. Αν υπάρξουν ε, λοιπόν εξαιρέσεις και από τις δύο πλευρές, τότε ο καταναλωτής απλά δεν ενημερώνεται. Ε, νομίζω πως ε, η οδηγία αυτή από ό,τι ακούσαμε κάνει τη ζωή μας πιο δύσκολη από τη πιο εύκολη. Βεβαίως γι' αυτό έχουμε τους εμπειρογνώμονες εδώ πέρα. Λοιπόν, ε, να υπενθυμίσω στου βουλευτέ που είναι ακόμα εδώ πέρα. Ε, κυρία Στάιλε, και ο κύριος Χατζημαρκάκης θέλει, θέλει να παρέμβει. Για να συνοψίσουμε βεβαίω, να συνοψίσει και η συγκέντρια και να μα πει το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα τρεις ε, θετικές ε, πτυχέ που θέλω να αναφέρω και που υποστηρίζω την κυρία Στάιλερ. Έχουμε τη συμπλήρωση των ορισμών, ειδικά για το θέμα στο άρθρο 2 επίσης επαρκείς ε, επαγγελματικές ε, γνώσεις ε, του ενδιάμεσου γιατί είναι περίπλοκα τα ασφαλιστικά προϊόντα θα πρέπει λοιπόν να επιτηρείται η εκπαίδευση του ενδιάμεσου από μια εθνική αρχή όπως ε, αναφέρεται στο άρθρο 8 επίσης χαιρετίζουμε την συμπλήρωση για την ε, παροχή επιπρόσθετων ε, πληροφοριών γιατί είναι όπως είπαμε περίπλοκες οι ασφάλειες και δεν μπορούμε να αναμένουμε από τον καταναλωτή να ξέρει ποιες είναι οι ερωτήσεις που πρέπει να θέσει. Και η κυρία Στάιλερ στο άρθρο 17 σωστά έχει κάνει κάποιες αλλαγές. Ένα σημείο κριτικής αφορά το πεδίο εφαρμογή, εκεί πέρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σε ποιον απευθύνεται τελικά η οδηγία. Είναι όλοι οι υπάλληλοι μόνο όσοι έχουν επαφή με τους πελάτες ή μόνο όσοι είναι ενδιάμεση. Αυτό δεν προκύπτει από την πρόταση. Με αυτές τις σύντομες παρατηρήσεις κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να ολοκληρώσω. Ωραία. Θα ήθελα και εγώ εκ μέρους της δικής μου πολιτικής ομάδας να πω ότι ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η ακρόαση. Και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που είπαν οι εμπειρογνώμονες για την ασφάλεια ό,τι αφορά την αναλογικότητα, γιατί είναι ευρύτερο το φάσμα των προϊόντων που καλύπτονται. Και είναι περίπλοκο το θέμα της παροχής πληροφοριών. Θα πρέπει να έχουμε ένα είδος, κάποιο τεστ αναλογικότητας γιατί είναι πολύ διαφορετικά τα είδη των ασφαλίσεων. Και άλλο το πεδίο των δραστηριοτήτων του κάθε διαμεσολαβητή. Οπότε το θέμα της ε, παροχής πληροφοριών ε, για τις αμοιβές σε τέτοιες περιπτώσεις είναι υπερβολικό. Θα πρέπει ε, επίση το θέμα των no claims bonuses να το λάβουμε υπόψη γιατί είναι περίπλοκο και δύσκολο. Επίσης, θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε στρέβλωση του ανταγωνισμού και να αποφύγουμε να ευνοήσουμε ένα μόνο κλάδο, μία μερίδα διαμεσολαβητών. Βέβαια, μερικές φορές υπάρχει η πρόσβαση μέσω ίντερνετ όπου κανείς χωρίς να καταβάλει καμία προσπάθεια μπορεί να διαφημίσει ένα προϊόν και υπάρχει και η επαφή με τον πελάτη γίνεται λίγο διαφορετικό εκεί το είδο τη δραστηριότητας και γι' αυτό και το θέμα των αποδοχών είναι περί, περίπλοκο και η παροχή πληροφοριών για αυτές ε, είναι επιμάχου θέμα. Ούτε θα πρέπει να είναι μεγάλη ε, η πληθώρα των πληροφοριών να καταιγίζεται ο καταναλωτής και να μην μπορεί να αποφασίσει. Θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της ανάγκης πληροφόρησης και το να μην είναι υπερβολικά εκτεταμένες ε, οι πληροφορίες. Η ευρεία χρήση του ίντερνετ για την πώληση προϊόντων επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και γίνονται προσφορές σε site ε, με τίτλους ε, συγκρίνεται τις αγορές» «Με συγκρίσεις τιμών». Σίγουρα γίνονται συγκρίσεις, αλλά δεν είναι αυθεντικές πάντα. Θα πρέπει να αν θέλουμε να κάνουμε τις συγκρίσεις, να καλύπτουν όλη την αγορά, γιατί υπάρχουν παραπλανητικές τέτοιες διαφημίσεις. Κυρία Στάιλερ, σίγουρα δεν είναι εύκολο το έργο σας για να προσπίσετε το συμφέρον των Ευρωπαίων καταναλωτών. Πείτε μας καταρχήν λίγα λόγια για το χρονοδιάγραμμα. Αν δεν κάνω λάθος, η προθεσμία των τροπολογιών είναι 22 Ιανουαρίου και όχι 7η Ιανουαρίου όπως αρχικά είχε αναφερθεί. Δεν ήμασταν βέβαια πολύ παρόντες, αλλά ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η ακρόαση, πολύ ποιοτικέ ε, οι ομιλίες και ακούσαμε τις ανησυχίες του κλάδου, των καταναλωτών, εκπροσώπων καταναλωτών και πόσο δύσκολο είναι να εξασφαλίσουμε σαφήνεια και ενάργεια για τέτοια θέματα. Φυσικά θέλουμε τη διαφάνεια, αλλά πώς ε, θα την εξασφαλίσουμε εξυπηρετώντας τον ε, καταναλωτή και βρίσκοντας και κάποια ισορροπία. Γιατί μιλήσαμε για τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων μορφών ασφαλιών ζωής και των υπόλοιπων ασφαλιών. Επίσης υπάρχουν ε, πολύ μεγάλοι παίκτες και πολύ μικρότερες εμβέλειες επιχειρήσεις. Δεν θα πρέπει να διακυβεύσουμε το καλό έργο που έχουμε κάνει υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επιβάλλοντα υπερβολικέ υπερβολικές υποχρεώσεις για αυτές, ό,τι αφορά ιδιαίτερα την παροχή των πληροφοριών. Πάντω, σε τελική ανάλυση, αυτό που θέλουμε είναι να εξασφαλίσουμε ενημέρωση των καταναλωτών, διαφάνεια στην παροχή πληροφοριών και μια συνεκτική πρόταση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συνεκτικότητα και με άλλες νομοθετικές προτάσεις που ταυτόχρονα δρομολογούνται. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει μια συνάφεια μεταξύ όλων αυτών των νομοθετικών προτάσεων. Στις τροπολογίες περιμένω τα σχόλια των σχεδόν εισηγητών και των υπόλοιπων μελών. Θα είναι σημαντικό να λάβω υπόψη και τα σχόλια των εμπειρογνωμόνων σε αυτά. Και μετά τη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών, γιατί ακόμη δεν έχει γίνει μια τέτοια, προσπαθήσαμε πριν τα Χριστούγεννα, τώρα θα ξαναοργανώσω συνάντηση των σκιωδών εισηγητών για να συνεννοηθούμε και να διευκρινίσουμε το θέμα των αρμοδιοτήτων μας με την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Θα το δούμε αυτό στη διάσκεψη των Προέδρων. Κανονικά θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και όχι διελκυνστίδα μεταξύ των Επιτροπών ΕΜΚΟ και ΕΚΟΝ. Αν δεν κάνω λάθο, οι μεταφράσει υπάρχουν αυτή τη στιγμή μόνο στα αγγλικά, γερμανικά και δανεικά. Θα πρέπει ε, να παρακολουθούμε και ταυτόχρονα φυσικά τις εξελίξεις των συζητήσεων στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Περιμένω τι τροπολογίε σα, αγαπητοί συνάδελφοι. Εξετάζω ήδη αυτές που έχουν υποβληθεί. Και ευχαριστώ για το χρόνο που αφιερώσατε στο θέμα αυτό. Και η Αγγέλικα... Ε, έκανε πολλές προσπάθειες. Η γραμματεία πραγματικά εργαστήκε άοκνα για να προωθηθεί η γνωμοδότηση αυτή. Ευχαριστώ όλους σας θερμά και ευχαριστώ φυσικά και τον Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντσέρη. Να επιβεβαιώσουμε λοιπόν 26 Ιανουαρίου προθεσμοί για τις τροπολογίες, θα δούμε τις συμβαστικές στις 20 ή 21 ή μετά ψηφίζουμε στις 4 Μαρτίου και η Επιτροπή Οικονομικών στις 26 Μαρτίου. Προφανώς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, αλλά λοιπόν, θα πρέπει να βιαστούμε και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να υπερασπίσουμε την Επιτροπή μας γιατί η ΕΚΟΝ ε, έχει θέσει πολύ σύντομο χρονοδιάγραμμα και αναμένουμε πως δεν θα αποφασιστεί τίποτα. Βεβαίω δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Θα προσπαθήσουμε να το καθυστερήσουμε, αλλά βλέπετε πόσο σοβαρά το παίρνουμε όσον αφορά την δική μας γνωμοδότηση. Και αυτά τα οποία είπατε βεβαίως θα τα μεταφέρω και στους ε, τέσσερις ε, ε, εμπειρογνωμονέ μας. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και σας ευχαριστούμε και για αυτά τα οποία μα είπατε. Την ε, Κομισιόν δεν την ακούσαμε, αλλά είχαμε πει πως θα ακούσουμε τους προϊστάμενους ε, στην επόμενη συνεδρίαση. Γι' αυτό δεν είχαμε σήμερα χρόνο για την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πάντως που ήρθατε. Ευχαριστώ και τους Ιερμηνείς ε, για τον λίγο παραπάνω χρόνο. Λύεται λοιπόν η συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίαση είναι 23 και 24 Ιανουαρίου για να ψηφίσουμε τέσσερα μεγάλα ε, θέματα. Αναμένω λοιπόν μια αίθουσα γεμάτη βουλευτές. Ε, εν τω μεταξύ εύχομαι καλή σας όρεξη. Ευχαριστώ πολύ.